Ladies and gentlemen, please Καθίστε παρακαλώ, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε με το τελευταίο κομμάτι των εργασιών μας αυτής της εβδομάδας, της Επιτροπής μας. Το πρώτο λοιπόν θέμα που θα συζητήσουμε Το πρώτο θέμα είναι η ρωσική στρατηγική επικοινωνίας και ο πληροφοριακός πόλεμος οι επιπτώσεις των πράξεων της Ρωσίας σε χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Είναι λοιπόν χαρά μου το ότι μου δίνετε ευκαιρία να καλωσορίσω τους ε, εξέχοντες ε, ομιλητές, Ζιλ Πόκμαν, Πόρτμαν, κάθεται εξ αριστερών μου, είναι επικεφαλής της ειδικής ομάδας East Stratcom και τον κύριο Πόρτμαν τον έχουμε συναντήσει ήδη αρκετές φορές κυρίως στην ομάδα των φίλων της Ουκρανίας, τις οποίες ηγείται ο κ. Στρεβίτσος. Έχουμε ακούσει μέχρι τώρα πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις εκ μέρους του και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε. Κατόπιν έχουμε την κυρία Βινέτα Μεκόνε του κέντρου του ΝΑΤΟ, του Κέντρου Αριστείας Στρατηγικών Επικοινωνιών του ΝΑΤΟ, που εντρεύει στη Ρήγα. Και ο τρίτος είναι ο κύριος Ρόμπερτ Πστέλ, που είναι επικεφαλής του Γραφείου Πληροφόρησης του ΝΑΤΟ στη Μόσχα. Υπάρχει τέτοιο γραφείο Έχω διαβάσει μία συνάντηση με τον κύριο Πστάλ και ο δημοσιογράφος περιγράφει τη δουλειά του ως τη χειρότερη δουλειά του κόσμου το να πρέπει κανείς ε, να ενημερώσει τη Μόσχα για τον ΝΑΤΟ. Αλλά, εν η δουλειά είναι και αυτή. Κυρίες και κύριοι, για σήμερα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα ημερήσια διάταξη. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Πόρτμαν, ο οποίος ε, θα μας ε, περιγράψει την Easter Stratcom και τις ε, επιπτώσεις από τη ρωσική στρατηγική Επικοινωνία στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως στους ανατολικούς μας εταίρους. Κύριε Πόρτμαν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους σας. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε σήμερα στη συνεδρίασή σας, εγώ θα καλύψω δύο θέματα. Πρώτον, ε, θα μιλήσω για τη φύση της πρόκλησης και δεύτερον, ε, θα σας εξηγήσω τι ακριβώς κάνουμε εγώ και οι συνεργάτες μου στην υπηρεσία, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Κοιτάξτε, εδώ δεν είναι μία ε, θεωρητική συζήτηση ή για κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, είναι για κάτι που συμβαίνει. Και δεν το λέω εγώ, το λένε και πάρα πολλοί άλλοι στη Μόσχα οι οποίοι ε, έχουν πράσει ε, επίσης την ίδια άποψη. Παραδείγματο χάρη έχουμε δει σχόλια τα τελευταία χρόνια στη Ρωσία για το ότι είναι απαραίτητο να γίνει ε, σύγκρουση πληροφοριακή για να μειωθεί το μαχητικό δυναμικό του αντιπάλου για να παραπλανηθούν οι ηγέτες ανατολικά ε, η Ρωσία είναι σε μόνιμο πόλεμο μόχωρης ε, στρατιωτικά μέσα και οι Υπουργοί Άμυνα ε, είπαν πέρυσι ότι η ενημέρωση γενικότερα είναι επίσης ένα όπλο των ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε μία απειλή την οποία να γνωρίζουν όλοι. Γι' αυτό λοιπόν το Μάρτιο του περασμένου έτους το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε για αυτό το θέμα και ανέθεσε τον ύπατο ε, εκπρόσωπο να συστήσει μια ομάδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, Εξωτερικής Δράσης και να καταθέσει ένα πρόγραμμα δράσης, το οποίο και έγινε, κατατέθηκε τον Ιούνιο. Ε, μετά συστήθηκε η δική μου ομάδα, η οποία λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, δηλαδή περίπου τέσσερις μήνες. Είμαστε μια ομάδα εννέα εκπροσώπων από τα κράτη-μέλη και τους θεσμούς. Οι περισσότεροι της ομάδας έχουν επαγγελματικό υπόβαθρο επικοινωνίας και γνωρίζουν και τη ρωσική γλώσσα. Και έχουμε τρεις στόχους. Ο πρώτος είναι να βελτιωθούμε στο να περιγράφουμε τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στην ε, ανατολική της γειτονία, πώς μπορεί να επικοινωνεί άμεσα με τους πολίτες επιτόπου. Το δεύτερο είναι να στηρίξουμε ε, τα πλουραλιστικά μέσα, κυρίως αυτά που λειτουργούν στα ρωσικά και το άλλο καθήκον μας είναι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση, αλλά επίσης και να ευαισθητοποιήσουμε για το πρόβλημα και εγώ θα μιλήσω γι' Η συνειδητοποίηση λοιπόν τριών πραγμάτων. Πρώτον, συνειδητοποίηση των τεχνικών ε, του πληροφοριακού πολέμου που είναι παραπλάνηση, ε, επιβράδυνση της λήψης αποφάσεων, υπονόμευση της αντικειμενικότητας. Βλέπουμε δηλαδή την τεχνική της συνεχούς ε, επανάληψης για το ποιος ε, είναι υπεύθυνο για αυτά που έγιναν στις 17 ε, Μαΐου. Ε, λέγεται ότι δεν υπήρχαν στρατιωτικά ρωσικά στρατεύματα στην Ουκρανία. Τα μέσα ενημέρωση προκαλούν την εντύπωση της αξιοπιστής, αλλά όλα αυτά που λένε είναι αβάσιμα. Μετά υπάρχει μια τεχνική όπου είτε αναφέρονται ε, λάθος ε, ρίσεις από ανθρώπους, λένε τελείως λάθος πράγματα ή ανακαλύπτουν, εφευρίσκουν κάποιον που υποτίθεται είτε ότι είπε κάτι και προκύπτουν μετά και ε, θεωρίες ε, Άρα δηλαδή ε, υπάρχει αμφιβολία και η αλήθεια ε, γίνεται πιο σχετική. Το άλλο που θέλουμε να, για το οποίο θέλουμε να προκαλέσουμε κάποια ευαισθησία είναι τα αφηγήματα. Υπάρχουν πολλά αφηγήματα. Υπάρχουν ε, αφηγήματα φενός και προπαγάνδα, ε, παραπλάνηση, ψέματα, πέσα το πώς θέλετε. Διαχωριστική μεταξύ, με, ανάμεσα στα δύο τα αφηγήματα δεν είναι απόλυτα λανθασμένα, είναι δηλαδή περισσότερο υποκειμενικά και όχι αντικειμενικά. Κατόπιν τούτου είναι πολύ δύσκολο να τα απορρίψει κανείς, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά αφηγήματα που υπονομεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τα οποία αυτά δηλαδή λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποτυχημένη, ότι θα καταρρεύσει, ε, λέγονται πολλά για την Ουκρανία, για τη Συρία και οφείλουμε όλα αυτά να τα αναγνωρίσουμε και να είμαστε έτοιμοι να τα αμφισβητήσουμε. Παράδειγμα, το αφήγημα ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα ε, της, του ηθικού μονοπωλίου ε, για το κληροδότημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μόνιμο αυτό. Ευαισθητοποίηση λοιπόν και για την παραπληροφόρηση, τα ψέματα και την προπαγάνδα. Βλέπουμε να υπάρχει τεράστια παραπληροφόρηση σε σχέση με την Ουκρανία. Υπάρχει αυτή η περίφημη ιστορία με το παιδί που σταυρώθηκε, που λένε άλλοι ότι δεν υπάρχουν ε, ε, Ρώσοι στρατιώτες στην Ουκρανία. 300 δημοσιογράφοι διακρίθηκαν με μετάλλια για το ότι διέδωσαν αυτή την πληροφορία. Το θέμα δεν είναι η παραπληροφόρηση στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά είναι παραπληροφόρηση που έρχεται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επηρεάζει και τα κράτη-μέλη. Ας πούμε την Ολλανδία του Άζοφ Πατάλιαν που Ουκρανός που υποτίθεται ότι θα έκανε τρομοκρατικές ενέργειες αν δεν ψήφιζαν σωστά οι Ολλανδοί. Αυτό ήταν ψέμα τελείως ή το λάθος του Λιντινάνκο στο Ηνωμένο Βασίλειο που είτε αυτοκτόνησε είτε δολοφονήθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου και οι αντιδράσεις για τις επιθέσεις της ε, πρωτοχρονιάς στην κολονία μια κοπέλα 13 χρονών που υποτίθεται απήχθη ε, και βιάστηκε και οι Γερμανοί δεν έκαναν τίποτα και αυτό αποδείχτηκε ψευτιά ψευτιά ολκής ε, Ας δούμε λοιπόν τι δείχνουν οι στιγμομετρήσεις. Οι μισοί Γάλλοι είπαν ότι φταίνε η... φταίει το Κίεβο. Επίσης, στην Ελλάδα οι περισσότεροι ε, είναι πιο κοντά στη Ρωσία από ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω, από ό,τι φαίνεται υπάρχει παραπληροφόρηση και δεν μπορεί να μας αρέσει αυτό. Έχουμε λοιπόν τρεις ε, βασικούς στόχους ε, στο πρόγραμμα δράσης που συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα τα αντιστρέψω γιατί μιλάμε για την παραπληροφόρηση. Θα μιλήσω λοιπόν πρώτα απ' όλα για τη δουλειά που γίνεται για την ε, παραπληροφόρηση. Εδώ η βασικότερη δουλειά είναι να εντοπίσουμε και να διαδώσουμε πληροφορίες για ψεύτικες ιστορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της. Και αυτό το κάνουμε μέσα από το Twitter, το θέμα Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την παραπληροφόρηση. Αυτό το επεξεργόζόμαστε στο διαδίκτυο και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που συμβάλλουν σε αυτό σε ε, εβδομαδιαία βάση. Μας επισημαίνουν ιστορίες που είναι λανθασμένες και η δική μας η δουλειά είναι να αναλύουμε ε, τη διάδοση της ε, παραπληροφόρησης Έχουμε ήδη λοιπόν ένα δίκτυο πολλών χιλιάδων ανθρώπων που διαβάζουν τις πληροφορίες που κυκλοφορούν στην Ευρώπη αλλά υπάρχει και περιορισμός για το πώς μπορούμε εμείς ε, να κυκλοφορούμε, να διαδίδουμε τις δικές μας πληροφορίες. Έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει έλλειψη ενδιαφερόμενων στα κράτη-μέλη. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ μπορεί να μας βοηθήσει το Κοινοβούλιο να ε, έρθει στο δικτυό μας και να μας βοηθάει να διαδίδουμε τις σωστές πληροφορίες. Το άλλο που κάνουμε είναι στηρίζουμε πλουραλιστικά μέσα στην περιοχή. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να συναγωνιστούμε τη χρηματοδότηση που προσφέρει το Κρεμλίνο στα μέσα του της ενημέρωσης. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία, αλλά ένα άρθρο στον Observer, EU Observer, λέει ότι τα λεφτά που δίνονται από το Κρεμλίνο είναι πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η Ρωσία εκπροσωπείται σε πάρα πολλές χώρες, υπάρχουν πολλά τρόλ που δεν μπορεί κανείς να τα εντοπίσει, χιλιάδες είναι. Εκατομμύρια ευρώ δαπανώνται επιτόπου σε ΜΚΟ. Ε, εμείς ε, δεν θα ε, εγκαταστήσουμε τηλεπτικό σταθμό, δεν πιστεύουμε ότι νομιμοποιούμε θα να κάνουμε κάτι τέτοιο, ούτε και τα λεφτά θα ήταν σωστά δαπανημένα. Οι χώρες, ε, η περιοχή της Βαλτικής και οι χώρες της ε, Ανατολικής Ευρώπης προσπαθούν να βελτιώσουν την εκπομπή ρωσικών και ρωσόφωνων εκπομπών γιατί υπάρχουν μειονότητες. Εν πάση εμείς συνεργαζόμαστε με φορείς όπως ε, το Ευρωπαϊκό Κληροδότημα για τη Δημοκρατία για να ε, έχουμε καλύτερη πηγή πληροφόρησης, ε, να έχουμε πλατφόρμες, την ανταλλαγή δημοσιογράφων έτσι ώστε να δίνουμε στη δημοσιογράφους όχι μόνο την εκπαίδευση αλλά και την πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης έτσι ώστε και αυτοί να είναι πιο ενημερωμένοι στα ρεπορτάζ τους. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι παρότι μιλάμε για παραπληροφόρηση, η ομάδα μου δουλεύει περισσότερο για θετική ενημέρωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η άλλη πλευρά της ε, παραπληροφόρησης. Την καταπολεμούμε, αλλά και πρέπει να αναλάβουμε την πληροφορία και να εξηγήσουμε τι ακριβώς κάνουμε. Και αυτό να το ανακοινώνουμε άμεσα. Παραδείγματος χάρη πρόσφατα παρουσιάσαμε ταινίε ε, για το φέλη του DCFTA στην Ουκρανία και για την απελευθέρωση των ε, θεωρήσεων, η πρόοδος που υπάρχει στη Γεωργία και την Ουκρανία ή φέτος μαζί με τις αντιπροσωπείς μας στην περιοχή ε, έχουμε μια εκστρατεία θετική ενημέρωσης για όλες τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Τελευταίο σημείο που θέλω να φέρω είναι το εξής. Δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, ενημερώσει σωστά ε, τους ρωσόφωνους ε, κατά το παρελθόν. Εμείς θέλουμε να το διορθώσουμε. Σας λέω όλοι στην ομάδα μας ξέρουν πολύ καλά ρώσικα, έχουν δουλέψει στη Ρωσία σε άλλες εκεί περιοχές και διασφαλίζουμε να έχουμε ομιλίες, δηλώσεις στα ρωσικά, να τα προβάλλουμε αυτά στους ρωσόφωνους δρομολογήσαμε ένα ιστότοπο στις 8 Φεβρουαρίου eeas.europa.eu ε, au το είναι ο ιστότοπος και αυτό είναι σημαντικό διότι καταρχήν ε, ένα μύθο ότι δηλαδή αν είναι κανείς ρωσόφωνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δήθεν σε αντιμετωπίζουν ως πολίτη δεύτερης κατηγορίας. Ψέματα. Εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι τα ρώσικα ε, είναι μια ε, αναγνωρισμένη γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς ε, θέλουμε να επικοινωνούμε άμεσα με τους ρωσόφωνους. Επίσης, από τότε που έχουμε φτιάξει την ιστοσελίδα μας, βλέπουμε πραγματικά εκατοντάδες εκθέσεις στα ρώσικα, θετικές αναφορές και επίσης ε, και ε, πολλές επισκέψεις στην ιστοσελίδα μας και αυτό δείχνει ότι πάνω από το 50% όλων των επισκέψεων στην ε, ιστοσελίδα μας έρχονται από όλο τον κόσμο και αυτό δείχνει ότι ανοίγει όρεξη και είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδίδει περισσότερο πληροφορίες στα ρώσικα. Εμεί θεωρώ ότι θα συμβάλλουμε σε όλα αυτά που γίνονται. Θα είμαστε ένα σημαντικό εταίρο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμεί ευχαριστούμε κύριε Πόρτμαν. Διαπιστώνουμε έτσι ότι το ΝΑΤΟ έχει προχωρήσει πάρα πολύ όσον αφορά την ε, ανείχνευση, επισήμανση, ε, αξιολόγηση ε, τι γίνεται με αυτού του είδους την απειλή για τις επικοινωνίες και έχουμε τον κύριο Στέλ μεταξύ των άλλων ε, προσκεκλημένων μας και τώρα ο κύριος Πιτσέλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ. Και εκτός από όλους τους άλλους λόγους νομίζω ότι οι δραστηριότητες και η πολιτική της ε, Ρωσίας μας δίνει ακόμα ένα κίνητρο ούτω ώστε να έχουμε αγαστή συνεργασία τα δύο θεσμικά όργανα. 4,5 χρόνια υπηρετούσα στην αντιπροσωπεία του ΝΑΤΟ στην ε, ε, Μόσχα. Και σήμερα ασχολούμαι με τα σχετικά θέματα, αλλά έχω υπηρετήσει και εκεί. Δεν θα σας εκπλήξει το ότι είμαι στο ίδιο με τον Giles, ε, αλλά να σας πω και δύο για το πρόβλημα να δούμε πώς έχει το τοπίο και στη συνέχεια να σας πω τι κάνουμε εμείς. Δεν νομίζω ότι θα βρείτε και πολλές διαφορές. Απλώς ε, κάποιες μικρές διαφορές οφείλονται στη διαφορά των δύο ε, οργανισμών. Έχουμε αυτή τη ε, πληροφόρηση, προπαγάνδα θέλετε, μοιάζουν πολύ αυτά από πλευρά Ρωσίας και αυτό είναι κάτι αδυσόπιτο, είναι κάτι συνολικό, σφαιρικό σαν δραστηριότητα γιατί εμπλέκει όλες τις κρατικές υπηρεσίες τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης που είναι υποέλεγχο γιατί ακόμα και τα μέλη του Ρεσκού Κοινοβουλίου ενεργά συμμετέχουν. Γενικά είναι μεγάλο πρόβλημα στη Ρωσία το ότι δεν υπάρχει ανεξαρτησία στα θεσμικά όργανα της κοινωνίας των πολιτών. Πρώτος ε, στόχος της προπαγάνδας βέβαια είναι ο ίδιος ο ρωσικός λαός. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Πολύ περιορισμένη προβληματική για αυτά τα θέματα στη Ρωσία. Αυτό έγινε και με την προσάρτηση της ε, Κρυμαίας. Ελάχιστα συζητήθηκαν. Πάρα πολύ λίγοι βουλευτές στην Τούμα. Κάτι πήγαν να πούν και μετά από μια ώρα σταμάτησε η συζήτηση, θεωρήθηκε χασίμο χρόνο. Οπότε θα πρέπει να καταλάβουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για μια πολιτική και από πλευρά μας δεν μιλούμε για τον ρωσικό λαό καθεαυτό. αυτό. Ό,τι λέμε για την προπαγάνδα δεν το λέμε για το ρωσικό λαό γιατί ο λαός είναι το πρώτο θύμα αυτής της προπαγάνδας. Οπότε ο στόχος είναι η δημιουργία μιας συγκεκριμένη εικόνας. Και η παράδοση λέει ότι το ΝΑΤΟ είναι ο πιο μεγάλος τους ο πρώτος στόχος της προπαγάνδας. Αλλά βέβαια εξαρτάται για ποια μέρα μιλάμε. Πολλέ πολλές φορές μπορεί να υπάρχει μια έκθεση που να αρέσει τη Μόσχα, άλλη φορά μπορεί να υπάρχει κάποια ε, επίκριση προς ε, τον ΟΗΕ. Τέλος πάντων υπάρχει εδώ κάποια ουδετερότητα, αλλά πάντως δεν εξαιρείται κανείς από το να είναι στόχος αυτής της πολιτικής. Να σας πω μια ακραία περίπτωση για πόσο μας έχουν ως στόχο πρόσφατα είναι κάποια εκδήλωση αρκετά προβεβλημένη. Και λίγε κάποια κιόσκια τα οποία θα κλείνανε, τα οποία θα ήταν κοντά στους σταθμούς του μετρό. Αυτό έγινε κρυπτό, ο κόσμος πάντως δεν ήταν ευχαριστημένος, το προβλήθηκε στον τοπικό τύπο αλλά είπανε ότι έπρεπε να καταστραφεί αυτό το και αλλιώς εκεί θα έπαιρνε τη θέση του τα τάγκς του ΝΑΤΟ. Να, κάτι τέτοια λένε, αλλά κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι κομμάτι του παιχνιδιού και είμαστε συνηθισμένοι. Τώρα όσον αφορά τις χώρες μας, όσον αφορά τις χώρες της ε, ανατολικής εταιρικής σχέσης. Το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέμε ότι προσπαθούν να μας φέρουν σε αντιπαράθεση με τη ΣΥΠΑ. Οι άλλες φορές προσπαθούν να υπονομεύσουν την αξιοπιστία. και έτσι να περικόψουν τις δυνατότητες ανάπτυξης και τις δυνατότητες εξωτερικής πολιτικής, εκτός αν η χώρα στόχος ευθυγραμμιστεί με τη Ρωσία. Δηλαδή, το θεματολογιό τους καλύπτει και την ε, υπόνομηση της αξιοπιστίας στο διεθνές σύστημα ασφαλείας. Να, κάτι πολύ σημαντικό από πλευρά στρατηγική. Χρησιμοποιούν λοιπόν διάφορου μύθου και κλισέ. Κλασικά πράγματα. Παρά το, το ότι έχει υπάρχει συνθήκη ε, με το άρθρο 10 που διέπει τον Άτο σε σχέση με την επέκτασή του. Λένε λοιπόν ψέματα σχετικά με αυτό. Ε, επίσης τα σχετικά με την Κρυμαία και τη Σεβαστούπολη. Αυτά δεν τα λένε κάποιοι ειδικοί. Προέρχονται ακριβώς από την κορυφή της πυραμίδας εκεί. Ας πούμε, έχουμε μια κρίση. Α, η κρίση του μεταναστευτικού, ένα ωραίο παράδειγμα. Και αμέσως η μηχανή αυτή αρχίζει να λειτουργεί και κάτι βγαίνει σε σχέση με την κρίση. Και φυσικά μαυρώνεται έτσι η Δύση, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα είπε το παράδειγμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ο Τζάλο, αυτή τη σχετική χειραγώγηση και το σχετικό αφήγημα. Και ο Μεντεβέντεφ πρόσφατα, ο Πρωθυπουργό, είπε ότι η Ρωσία είναι μια φιλιρινική χώρα. Και η απόδειξη είναι ότι όταν η Τουρκία κατέριψε το ρωσικό μαχητικό δεν απαντήσαμε αναλαμβάνοντας στατική δράση. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έξυπνο γιατί βεβαίω κατερίθεται το αεροπλάνο γιατί επανειλημμένα παρεμβεί στον εναερίο χώρο μιας ε, κυριαρχής Χώρα που είναι και μέλο του ΝΑΤΟ. Όμως ε, αυτό είναι ένα παράδειγμα για το τι κάνουν ούτω ώστε να προβάλλουν τη χώρα τους ω φιλιρινική ακόμα ε, και όταν προβάλλουν τέτοια παραδείγματα χτύπητα κάθε μέρα επίσης ακούμε για τις επαφές ΝΑΤΟ και Ρωσία αυτό το περίφημο Συμβούλιο Επαφής που υπάρχει ε, όπου είναι βήμα διαλόγου αλλά βέβαια, έτσι όπω προβάλλουμε τη λειτουργία του Συμβουλίου, πάντα προβάλλουμε το τι κάνουν εκείνοι. Κάποια θυμότητα τη αρχή. Πρώτα απ' όλα, εμεί δεν κάνουμε προπαγάνδα. Επομένω, δεν θα πολεμήσουμε την προπαγάνδα με προπαγάνδα. Αυτό θα ήταν κατά των αρχών μα. δεν θα απέδιδε, αλλά δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Ούτε επίση είναι μία σου και μία μου η αντίδρασή μα, η νοοτροπία μα γιατί αυτό θέλουμε δεν είναι αξιοπρεπές γιατί πολλά από αυτά τα επιχειρήματα είναι τέτοιο επίπεδο που ούτε να τα επαναλάβω να σας τα πω δεν τολμώ οπότε δεν θα γινόταν κάτι τέτοιο από την άλλη μεριά γιατί έχουμε όλους αυτούς τους ε, αναλυθείς ισχυρισμού, τους μύθους κλπ. κλπ. οπότε γι' αυτό σας λέω ότι δεν ανταποκρινόμαστε, δεν απαντάμε με παρόμοιους τρόπους, με μύθους και παραπληροφόρηση. Πέραν αυτού βεβαίως και δίνεται κάποια απάντηση. Είναι θέμα αυτοάμυνας. και θα πρέπει τα πιο κατάφορα, τα πιο χτυπητά που λένε πρέπει να τα απαντήσουν. Πάντως, εμείς δεν εκφραζόμαστε με έλλειψη σεβασμού για τη Ρωσία, για το ρωσικό λαό. Δεν κάνουμε αυτό που κάνουν εκείνοι προς εμάς. Και σας καλώ να διαβάσετε ε, κάποιες δηλώσεις του υπέξ της ε, Ρωσίας. όπου τακτικά, εβδομαδία σε εβδομαδία βάση, προσβάλλει και θίγει. Οπότε αυτό επίσης που βαρύνει πολύ είναι όταν κανείς ε, κατονομάζει στα πλαίσια της ε, χειραγώγης, οπότε και εμείς θα πρέπει να απαντούμε ότι πρόκειται για κάτι αναλυθές, πρόκειται για χειραγώγηση, ότι πρόκειται για προπαγάνδα, αλλά θα πρέπει κανείς να κατονομάζει τις ενέργειες. Και μιλάμε τώρα για τους συμμάχους, για τις διεθνείς, τους οργανισμούς, οπότε Υπάρχουν δημοσιεύσεις, υπάρχουν websites ε, για την διόρθωση των λεγόμενων και μέσω του Twitter προσπαθούμε να στείλουμε το μήνυμα. και στα ρωσικά εν και υπάρχει και γραφείο ενημέρωση στην ε, Μόσχα. Επίσης έχουμε και άλλα μέσα απάντησης όταν δηλαδή μπορούμε προβάλλουμε κάποιες εικόνες από τον δορυφόρο ή τους δορυφόρους για να προβάλλουμε την στρατιωτική δράση των Ρώσων στην Ουκρανία. Προσπαθούμε όλα αυτά να τα κάνουμε με την μέγιστη την αντιδιαφάνεια και ό,τι κάνουμε το επόμενο εξάμεινο όλα αυτά υπάρχουν στο website. Επίσης ε, οργανώνουμε συνεντεύξεις τύπου ε, και για τους Ρώσους δημοσιογράφους. Να πως ε, απαντούμε. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό αυτό που κάνουμε. Και με διάφορους τρόπους. Ας πω ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δίνει 200 συνέντευξεις το χρόνο και έχουμε επαφέ με τα μέσα ενημέρωση τακτικά και όχι μόνο με τα ΜΜΕ. Άρα προσπαθούμε κατά κάποιο τρόπο να βοηθήσουν. Είναι θέμα βέβαια και οικονομικών πόρων ε, για τη βοήθεια αυτή προς τους εταίρους μας, για Γεωργία, για Ουκρανία, για να μπορέσουμε να τους θωρακίσουμε κατά κάποιο τρόπο, να τους θωρακίσουμε καλύτερα, τους καλούμε σε σεμινάρια. Αν θέλουν, τους συμβουλεύουμε. Και έτσι να έχουν συστήματα πιο αποδοτικά. Αλλά θεωρούμε ότι το βασικό και η καλύτερη βοήθεια προς αυτές τις χώρες για να θωρακιστούν από την παραπληροφόρηση είναι να τις βοηθήσουμε όσον αφορά το μέτωπο των μεταρρυθμίσεων. Γιατί η Ρωσία δεν θέλει αυτές οι χώρες να κάνουν τις μεταρρυθμίσεις γιατί αυτό υπονομεύει τη ρητορική, την ρωσική. Άρα δεν πηγαίνουν καλά αυτές οι χώρες, δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν. Οπότε βοηθώντας τους ε, εταίρους μας ακριβώς και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πολύ περισσότερο από ότι το ΝΑΤΟ. Άρα αυτό το θετικό θεματολόγιο είναι πολύ σημαντικό. δεν θέλω να διαφωνήσω με τον Τζέλης, απλώς ε, θέλω να σας πω τώρα στο τέλος της εισήγησής μου ότι όπως είπε ο Τζάιλς αυτού του είδους οι ρωσικές προσπάθειες εν μέρη πιάνουν τόπο. Δημιουργούν αυτή την γκρίζα περιοχή, ούτε αλήθεια ούτε αναλήθεια. Α, βλέπετε το Russia Today, καλή ξέρω εγώ πέντε προσκεκλημένους οι οποίοι βλέπουν τις απόψεις ε, και που λένε κάτι περίεργα πράγματα σαν να ήταν η ναι, Τέλος πάντων η αλήθεια είναι κάπου στη μέση σε σχέση με τι συμβαίνει. Αλλά έχουμε και το τι γίνεται με τα ΜΜΕ των χωρών του ΝΑΤΟ. Τις απόψου προφανώς για τη ρωσική πολιτική και μόνο 26% από αυτά τα Ε. είναι υπέρ ενώ 62% είναι κατά. Δηλαδή η ρωσική πολιτική έχει χάσει πάρα πολύ σε αξιοπιστία. Δεν υπάρχει σχέση εμπιστοσύνη προς αυτήν. Και έχουν ξοδευτεί πάρα πολλά χρήματα για να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα της προπαγάνδας της χώρας μας. Άρα θα ήταν ε, αυταπάτη να πει κανεί ότι καταφέρανε οι Ρώσοι να αποσπάσουν την πόσα αποτελέσματα. Αλλά τέλο πάντων υπάρχουν κάποια ανησυχητικά σημάδια τελευταία ότι δηλαδή το σημερινό αφήγημα, το σημερινό μήνυμα από τα ρωσικά μέσα είναι το ότι περιγράφουν τη χώρα σε κατάσταση πολέμου προς τον υπόλοιπο κόσμο, οικονομικό πόλεμο ή κανονικό πόλεμο. Πολύ επικίνδυνο αυτό, γιατί είναι χώρα που στρατιωτικοποιείται σύμφωνα με όλα αυτά Υπάρχουν γυμνάσια από πλευρά των ενόπλων δυνάμεων σχεδόν κάθε μέρα κλπ. Οπότε τέτοιου είδου μήνυμα και αφήγημα ενισχύει αυτή την ήδη επικίνδυνη τάση. Αυτό μας ενισχύει κάπως. Και σας ευχαριστώ. Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Πινέτα Μεκόνε από το κέντρο αριστείας ε, του ΝΑΤΟ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα. Με τιμά ε, παρουσία μου απόψε, σήμερα το πρωί μάλλον μαζί σας. Το κέντρο αριστείας πρόσφατα ιδρύθηκε αλλά ήδη έχουμε επεξεργαστεί πολύ το σημερινό θέμα. Θα ξεκινήσω με κάποιες διαφάνειες για το κέντρο. Η ιδέα είναι να παρέχει συνεισφορά στην βελτίωση των στρατιωτικών ε, δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ. Διεξάγουμε έρευνες, στηρίζουμε την εκπαίδευση και κατάρτιση για τις στρατηγικές επικοινωνίες, ε, αναπτύσσουμε έννοιες, ε, δόγματα, στηρίζουμε επίσης τις διάφορες ασκήσεις και γνώσια του ΝΑΤΟ δεν είναι βέβαια ένας οργανισμός ε, του ΝΑΤΟ, είναι ένα γραφείο που στηρίζει ε, τη δυνατότητα στρατηγικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ. Το κέντρο αυτό αρχικά ιδρύθηκε από τη Λετωνία. Εν συνεχεία προσχώρησαν έξι χώρες, επομένως ε, δημιουργήθηκε ως Διεθνής Οργανισμός και από 1η Σεπτεμβρίου πιστοποιήθηκε ως, ε, ως ένα κέντρο αριστείας του ΝΑΤΟ. Θα ήθελα όμως να παραλείψω την επόμενη διαβάνεια. Νομίζω ότι τα προανέφερα τα σχετικά ο συνάδελφος ε, τώρα. Που εστιάζουμε μέχρι στιγμή στο κέντρο μας, ε, στις ευρυδικές μορφές ε, πολέμου, στην κοινωνική στρατηγική της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, πληροφορίες για τον ΤΑΕΣ, στρατηγικές επικοινωνίες με τους συμμάχους μας κτλ. αρκετές είναι δράσιμο στο τομέα ε, της διεθνούς προπαγάνδας. Επίσης ε, εξετάζουμε και την έρευνα γιατί θέλουμε να δούμε αν όλες ε, αυτές οι στρατηγικές ευθυγραμμίζονται και συμπληρώνονται για να δούμε τι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Τώρα έρχομαι στο θέμα μας. Η πρώτη έρευνά μας ήταν για την Ουκρανία ακριβώς και έγινε στα τέλη του 2014, αρχές 2015. Ποια ήταν τα πορίσματα. Ήδη από τότε διαπιστώσαμε ότι η νημερωτική εκστρατεία και οι σχετικές αστικές δράσεις της Ρωσία, Ρωσίας ε, αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά μιας νέας μορφής ε, πολέμου όπως έχει πει και ο αρχηγός ε, Γεθά Γεράσοφ ένα χρόνο πριν ε, Γερασίμοφ, συγγνώμη, πριν από ε, την κρίση στην Ουκρανία. Και θα πω πιο πολλά για το δόγμα του στις επόμενες διαφάνειες. Φαίνεται ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες πραγματικότητες όπου προσλαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη σημασία από τη στρατιωτική ισχύ η επικοινωνιακή στρατηγική Υπάρχει έλεγχο στο μέσο μα και σε ενημέρωση στη Ρωσία και αυτό είναι πολύ σημαντικό και στην κρίση τη Ουκρανία. Ποιο είναι ο δυνατό ρόλο των συμπατρετών και των ε, κοινοτήτων τη Διασποράς. Αυτό πρέπει να είναι πολύ, ε, ένα θέμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη και στι χώρε τη όμορφη με τη Ρωσία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αναφέρθηκε και από τον συνάδελφο ότι υπάρχει και μια άλλη όψη του νομίσματος τη κοινωνική στρατηγική της Ρωσίας ή τι ότι με πολλή επιτυχία επηρεάζει το ακροατήριο και ε, το ρωσικό πληθυσμό και τη διασπορά. Αλλά είναι και κάπως αντιπαραγωγική αυτή η στρατηγική γιατί αποξενώνει άλλα ακροατήρια, Ουκρανία, ΝΑΤΟ, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η τακτική ε, είναι παρελκυστική ε, για την διασπορά και ψευδών πληροφοριών, δίνουν διαφορετικές βερσιών κάποιων γεγονότων, όλα αυτά πολύ γρήγορα ε, διαβιβάζονται, αλλά αυτό απαιτεί πολύ μεγάλη προσπάθεια, χρόνο, χρήμα. Και ε, η Ουκρανική κυβέρνηση, το ΝΑΤΟ και τα ανεξάρτητα μέσα, ανεξάρτητα εμπειρογνώμονες και οι πολίτες ε, χρειάζονται επίση πάρα πολύ χρόνο για να τα μελετήσουν και να ε, ανασκευάσουν όλα αυτά. Να σας δείξω τώρα κάποια ζητήματα. Τα βλέπετε όλα στην ιστοσελίδα μας και δεν θέλω να ε, μακρηγορήσω. Λοιπόν, πρώτη έρευνα στη διαφάνεια αναλύει την πολιτική ρητορική το πολιτικό περιεχόμενο, τα αφηγήματα σε διάφορες οπτικοακουστικές πλατφόρμες από τότε που ξεκίνησε η κρίση στην ε, Ουκρανία και εντοπίζει τις τεχνικές, ε, τις χειριστικές που χρησιμοποιεί η Ρωσία στην ε, επικοινωνιακή της στρατηγική. Με την δεύτερη έρευνα προσπαθήσαμε να δούμε πώς... Όχι, δεν είναι σωστή διαφάνεια αυτή. Μια πίσω. Την πρώτη σας την ανέφερα. Αναλύουμε λοιπόν πολιτικό περιεχόμενο, πολιτική ρητορική. Και η Δεύτερη, νέα έρευνα πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε, δείχνει πω μέσω των μασικών μέσα επικοινωνία επηρεάζει τι ευρωατλαντικέ αξίε και επανακαθορίζει την αρχή δημοκρατίας, ελευθερίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εμπιστοσύνη στους η ε, Ρωσία με την επικοινωνική στρατηγική και αυτά θα τα πω και στην τελευταία μου διαφάνεια. Ήδη προανέφερα τον ε, στρατηγό Γεράσιμοφ. Υβριδικός πόλεμος είπα. Αυτό είναι το δόγμα του Γεράσιμοφ και αυτό το έγγραφο σας δείχνει ακριβώς τα χαρακτηριστικά αυτά τα ε, στοιχεία του δόγματος. Δείχνει λοιπόν ότι οι ε, πληροφορίες έχουν πλέον στρατηγική σημασία και για την ασφάλεια. 21ος αιώνας κατά τον Γερασίμοφ έχει την τάση ε, κάπως να μην ξεκάθαρο η κατάσταση πολέμου, η κατάσταση ειρήνης. Θα μπορούσε δηλαδή μέσα σε μήνες ή και ημέρες ακόμα ένα κράτος που φαίνεται να είναι ε, σε ευμάρια να μετατραπεί σε ένα θέατρο ε, αναταραχής και παρέμβασης. Αυτό γίνεται με τη μετατόπιση διαφόρων εφαρμοσμένων μεθόδων χρησιμοποιούνται πια περισσότερο από μη στρατιωτικά ε, διάφορα μέσα, οικονομικά ε, κτλ. Και έτσι διανοίγονται ασυμμετρικές δυνατότητες. Οπότε τα στρατιωτικά μέσα απλά συμπληρώνουν αυτές τις προσπάθειες. Βλέπουμε από την αρχή της ε, ε, σύγκρουσης που δεν είναι καν ορατή ε, να χρησιμοποιούνται όλα αυτά τα, τα μέσα, όλες αυτές οι μέθοδοι. Βλέπετε στο διάγραμμα ότι θα πρέπει να προσέχουμε τι γίνεται στις επικοινωνίες. Εμείς θα πρέπει να εμένουμε στα στρατηγικά μας μηνύματα και να παρακολουθούμε την κατάσταση όσο εξελίσσεται. έχουμε διαμετρικά αντίθετα μηνύματα και αυτά χρησιμοποιούνται για δύο διαφορετικά ακροατήρια. Για ποιο λόγο. Διότι είναι διαφορετική συμπεριφορά που αναμένεται από τα δύο ακροατήρια. Το ίδιο μήνυμα, εντελώς αντίθετο ε, στην Ουκρανία και εντελώς αντίθετο στη ρωσική γλώσσα. The next slide. The next slide is already... Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε αυτή την πολύ ατυχή περίπτωση του Σλοβιάνσκα αναφέρθηκε. Υπήρξαν και συνεντεύξεις από κατοίκους του Σλοβιάνσκ και άτομα που ζούσαν κοντά στην κεντρική ε, πλατεία, αυτές οι μπαμπούσκας που συνήθως δεν ξέρουν τίποτα ε, και που δεν πήραν είδηση ακόμη και αυτές που ζουν εκεί στο Σιλοβιάνσκ, δεν πήραν είδηση για αυτό το συμβάν. Γιατί σας το λέω. Γιατί θέλω να στρέψω την προσοχή σας στην ε, εκδοχή ε, της ιστορίας από τις μπάμπουσκας. Για τους πιο πολλούς έχει συμβεί, γιατί δεν έχει ε, γίνει γνωστή άλλη βερσιόν. Δηλαδή αυτό που λένε οι γιαγιάδες δεν είναι γνωστό, άρα πολλοί έχουν μείνει με λάθος εντυπώσεις. Τι θέλει να πετύχει λοιπόν η Ρωσία, όπως σας είπα, χρησιμοποιεί αυτά τα διαφορετικά ακόμη και αντίστοιχα μηνύματα ανάλογα με το ακροατήριο στις ε, χώρες που στοχεύει αναζητεί να επιβάλλει τη σύγχυση, την παραπληροφόρηση, να απογοητεύσει, τη να αποδιοργανώσει την κοινωνία, να διαβάλει και να διαβρώσει τη δημόσια υποστήριξη προς το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την καθυστέρηση επίσης των ε, μεταρρυθμίσεων επιδιώκει, όπως και να στηρίξει κάποιες αντιπολιτευτικές ή ακραίες δυνάμεις, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει όταν της δοθεί ευκαιρία. Να, δια... να καθυστερήσει τη διαδικασία λήψη αποφάσεων ή να την αποπροσανατολίσει. Επιδιώκει να διαιρέσει την κοινωνία όχι μόνο με βάση την εθνικότητα. Τώρα, αυτό στι άλλε χώρε. Στη Ρωσία, η στόχη αυτή τη επικοινωνική στρατηγική με, την, ε, με τον περιορισμό στην πρόσβαση σε άλλες πηγές πληροφοριών μέχρι και εντός συνόρων, ποιος είναι ο στόχος. Μια κοινωνία που δεν έχει σωστή ενημέρωση, επαναπροσδιορισμός των δημοκρατικών αξιών, ένας άλλος στόχος, θύμος της αντιπολίτευσης και έλεγχος των μέσων που ήδη βέβαια τον έχει κυβέρνηση τον έλεγχο των μέσων ενημέρωση. Τώρα, ποια είναι τα στρατηγικά κέρδη, ποια είναι τα στρατηγικά ωφέλη τη Ρωσία. με αυτή την ε, χρησιμοποίηση τη επικοινωνική στρατηγική ω όπλου είναι ο επαναπροσδιορισμός των ευρωατλαντικών αξιών. Η υπονόμευση της τρέχουσας τάξης ασφαλείας στον κόσμο και ιδίως στην Ευρώπη. Άλλος στόχος είναι Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία να μην μπορέσουν να ενταχθούν ε, στην ευρωατλαντική συμμαχία. Προσπαθεί να δημιουργήσει αμφιβολίες, δυσπιστία, καχυποψία σε σχέση με οποιαδήποτε πληροφορία. Άρα οι χώρες αυτές ουσιαστικά δεν μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους ε, κατοίκους των χωρών. Στο αυτό το πρώτο σημείο που είναι ο παναπροσδιορισμός των ευρωπαϊκών αξιών. Η Ρωσία αμφισβητεί την ε, αξιοπιστία των εθνών οργανισμών και το προϊόν του έργου τους. Δηλαδή όλοι μπορούν να αφισβητούν ε, και άλλες κυβερνήσεις αλλά και τη δική τους κυβέρνηση. Οι δηλώσει, η ερμηνεία των διεθνών συμφωνιών κατά τη Ρωσία και πάντα από τις δυτικές χώρες και τους συμμάχους τους έρχονται σε αντίφαση με αυτές τις συμφωνίες. Επίσης η ηθική υπεροχή της Ρωσίας, ε, δηλαδή ότι τελικά μια χώρα μπορεί να είναι ανώτερη από κάποιες άλλες. Είναι ένα μήνυμα επίσης, ένα αφήγημα. Και ο ρόλος της Εκκλησίας προβάλλεται ιδιαίτερα λέει ότι η Ευρώπη δεν είναι ενωμένη, η Δύση δεν είναι ενωμένη, ούτε και στις απόψεις τους, η Δυτική είναι ενωμένη. Επηρεάζονται τα μέσα, έχουν καθεί αξίες, προέχουν οικονομικά συμφέροντα, η ελεύθερη αγορά είναι μειονέκτημα και δείχνει την αποτυχία του δημοκρατικού συστήματος διακυβέρνησης. Οι τοπικοί αγρότες πλήττονται, δεν προστατεύονται προστατεύονται από χαμηλής ποιότητας ε, προϊόντα. Αλλά αν όμω υπάρχει ελεύθερη αγορά στη Ρωσία, θα υπάρξει διαφοροποίηση με προϊόντα από Αφρική, Λατινική Αμερική και Ασία για τη Ρωσία. Αυτά είναι τα πορίσματα. Αφού αναλύσαμε τέσσερις συγκεκριμένε υποθέσεις, τη Συμφωνία Μινσκ 2, τι ε, αντικυρώσει ε, από τα αντίπεινα δηλαδή από την ε, Ρωσία σε εξελίξει της 17ης Μάη και οι αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας. Επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπετε την ανάλυση των αφηγημάτων της Ρωσίας προς το δυτικό ακροατήριο και το ρωσόφωνο ακροατήριο. Εδώ μπορούμε να δούμε ποιες τεχνικές χρησιμοποιεί η Ρωσία πώς μπορεί να επαναπροσδιορίσει και να επανακαθορίσει με αυτή τη στρατηγική της τις ευρωατλαντικές Αυτά και σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουν ζητήσει πάρα πολύ το λόγο. Πρώτα απ' όλους ο κύριος Γκάλα. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας ε, είπατε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχει κανείς έτσι μια γενική εικόνα για το περί τίνος πρόκειται. Και πρέπει να σας πω ότι είμαι ευγνώμων ε, που έχουμε αρχίσει να αντιδρούμε. Νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι να ευαισθητοποιήσουμε την δημοκρατική κοινή γνώμη ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Να γνωρίζουν όλοι ότι υπάρχει αυτός ο πόλεμος προπαγάνδας. Γιατί η δική μας η ανοιχτή κοινωνία επιζητά περισσότερο την αρμονία, την ισορροπία, το συμβασμό και η αντίδραση των ανθρώπων είναι ε, κάπου στη μέση τα αλήθεια. Και αυτό αρκεί στη ρωσική πλευρά. Δηλαδή να μπαίνουν όλα στην ε, ίδια ζυγαριά, το τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα, τι είναι μισοαλήθεια, μισοψέμα. Ε, αν ισχύει αυτό τότε κερδίζει η ρωσική πλευρά. Και βλέπουμε τις ε, επιπτώσεις. Έχουν περιγραφεί στη επιπτώσεις στη Δυτική Ευρώπη και νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να αντιδρούμε. Ακόμα και αν γνωρίζουμε ότι εντωμεταξύ βλέπουμε ότι υπάρχει χρηματοδότηση των ε, ακραίων δεξιών κομμάτων. Ε, το ερώτημά μου είναι το εξής. Λόγω των ε, περιορισμένων πόρων που υπάρχουν ε, και στους δύο φορείς, μήπως έχει νόημα αυτές οι δραστηριότητες να συντονίζονται. Κατά την άποψή μου δεν θα πρέπει να εργαζόμαστε παράλληλα, αλλά να συνενώσουμε τις δυνατότητές μας και με τον τρόπο αυτό να είμαστε αποτελεσματικότεροι. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξή, ε, που εντάξει δεν θα το απαντήσετε εσείς, ε, θέλει χρήση πολιτικής απάντησης, Είναι όμως το εξή. Χρειαζόμαστε ρωσική τηλεόραση στη Δυτική Ευρώπη που να μην ε, είναι προπαγανδιστική. Υπάρχουν ε, κάποιες ε, προσπάθειες από εκείνους τους Ρώσους που έρχονται στη Δυτική Ευρώπη να δημιουργήσουν κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο εμείς πρέπει να το χρηματοδοτήσουμε. Και άλλο ένα παράδειγμα. Ας πούμε, στη ρωσική τηλεόραση έτρεχε μία δήλωση την οποία όμω ε, την είδαν και 11 εκατομμύρια ρωσόφωνοι στη Δυτική Ευρώπη και στο Ισραήλ. Στη ρωσική λοιπόν ε, τηλεόραση αναφερόταν ότι οι πρόσφυγες είναι επικίνδυνοι για την υγεία σας. Είναι βακτηριολογική βόμβα, δεν ε, μας απειλούν μόνο οι τρομοκράτες, εκατομμύρια Ευρωπαίων ε, θα μπορούσαν να πεθάνουν από μολυσματικές ασθένειες. Αυτό λοιπόν ήρθε από τη ρωσική τηλεόραση ε, και δημιούργησε μια συγκεκριμένη κατάσταση στη Δυτική Ευρώπη. Αυτά λοιπόν τα απίστευτα είναι ένα από τα πολλά. Γι' αυτό πρέπει να εξοπλιστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε, αλλά χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό και μεγαλύτερες δυνατότητες. Ο κύριος Πασκού. Ε, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ε, θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή ΣΕΝΤΕ για την ε, οργάνωση της χθεσινής και της σημερινής πολύ ενδιαφέρουσας συνεδρίασης. Όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε είναι πολύ πολιτικά και όσο πιο πολύ συναντιόμαστε και ανταλλάσσουμε απόψεις τόσο το καλύτερα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι κάποια στιγμή ξέρετε πρέπει και εγώ να φύγω γιατί πρέπει να προλάβω το αεροπλάνο μου. Και αυτό δεν είναι παραπληροφόρηση. Πάντως, κοιτάξτε, έτσι σε γενικές γραμμές ε, έχουμε δύο πλευρές. Έχουμε τις ηγετικές φυσιογνωμίες και αφενός την κοινή γνώμη και στη Ρωσία και στη Δύση. Και υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούμε όχι. Ξέρετε, η Δύση είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της Ρωσίας. Αυτό δεν είναι μυστικό και νομίζω ότι γνωρίζετε αυτή η ιδέα ότι η Ρωσία δέχεται επιθέσεις, ότι είναι εγκλωβισμένη έχει προεκτάσει, Δηλαδή, στη Ρωσία μπορεί ας ο ηγέτη να πει ότι ξεχάσετε τη δημοκρατία και τα συναπή, πρέπει να σώσουμε τη χώρα, παραδείγματο χάρη. Και έτσι βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο το οποίο επιθυμούν να μεταφέρουν στους πολίτες τους. Και θέλω να σας πω το εξής. Αν πάρουμε τις ε, πολιτικές φυσιογνωμίες και την κοινή γνώμη θα πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας εδώ στη Δύση, στην κοινή γνώμη στη Δύση. Γιατί εδώ δεν μπορεί κανείς ε, να πείσει τους ε, ηγέτες ότι κάνουν λάθος, γιατί θέλουν να κάνουν λάθος. Υπάρχει ας πούμε η αντιπυραυλική άμυνα. Εγώ έρχομαι από τη Ρουμανία και Οι Ρώσοι πολλές φορές ε, μας ε, προσάπτουν πράγματα. Τους λέμε ότι δεν είναι έτσι, αλλά αυτοί συνεχίζουν να ισχυρίζονται ότι πρόκειται για... Ε, είναι στρατηγική τους. Δεν θέλουν να πιστούν. Και κάτι άλλο, σε παρένθεση. Εμείς πάντα ενδιαφερόμαστε όταν επενδύουμε κάτι τι θα αποκομίσουμε. Αλλά η Ρώση δεν ενδιαφέρεται και γι' αυτό ε, ακόμα και αν πετάνε τα λεπτά από το παράθυρο δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει να σπείρουν ε, και στρατιώτες όλο τον κόσμο και να σφαγιάζονται. Δεν τους νοιάζει. Γιατί μπορούν να το κάνουν αυτό και στο τέλος ε, πιστεύουν ή μπορεί και να γίνει να επικρατήσουν. Αυτά για την ηγεσία στη Ρωσία. Τώρα, κοινή γνώμη, οι πολίτες στη Ρωσία είναι δύσκολο να επηρεαστούν για πάρα πολλούς λόγους. Και εγώ ανησυχώ για ένα πράγμα που είναι στρατηγικής φύσεως, είναι σημαντικό και πρέπει κάπως να αντιμετωπιστεί. Έχουμε να κάνουμε με μια νέα γένεια Ρώσων, οι οποίοι ε, μεγάλωσαν, ανατράφηκαν με μίσος εναντί της δύση. Αυτοί λοιπόν ε, θα φέρουν σε όλη τη ζωή αυτή την κατήχηση και εδώ ξέρετε εγώ έχω πρόβλημα γιατί αυτοί είναι οι νέοι οι οποίοι ε, θα πρέπει ε, να γνωρίσουν κάπως ε, τη σύγχρονη επικοινωνία. Τι κάνουν όμως, καταπίνουν τα ψέματα που τους πετάνε κατάμουτρα με μεγάλη ευκολία. Έτσι λοιπόν η Δύση, εκεί, εδώ στη Δύση θα πρέπει να προστατευτούμε, εδώ θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την προπαγάνδα αναφέρατε κάτι ε, για το τι κάνουν ή έκαναν, ας πούμε, για να πειράσουν τους Ολλανδούς στο δημοψήφισμα και αποδείχτηκε όλα αυτά ήταν ψέματα. Τώρα, οι Ολλανδοί ενημερώθηκαν γι' αυτό, γιατί αν το ξέρουν μόνο οι πολιτικοί ε, και δεν το έμαθαν οι πολίτες, τότε πέτυχαν το στόχο τους τι σημασία έχει που ξέρουμε εμείς ότι ήταν ψέμα. Το ψέμα πέτυχε το στόχο του. Νομίζω λοιπόν ότι κατόπιν τούτου θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας περισσότερο εδώ ε, στην κοινή γνώμη στη Δύση, όσο και αν είναι παράδοξο. Δεν λέω ότι πρέπει να ξεχάσουμε πλήρως τους Ρώσους, αλλά θα πρέπει να μας απασχολεί περισσότερο η νέα γενιά. Ορισμένα πράγματα μπορούν να γίνουν και στη Ρωσία, ε, αλλά σε μεγάλο βαθμό θεωρώ ότι εμείς και η δική μας η κοινή γνώμη ε, εδώ θα πρέπει να στραφεί η προσοχή. Η δική μας η πολιτική θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν περισσότερο όλα αυτά, γιατί μερικές φορές οι πολιτικοί μας ε, δεν τα προσέχουν. Εσείς τα προσέχετε γιατί είσαστε τεχνοκράτες. Τώρα πόσο μπορείτε να πείσετε τους πολιτικούς ότι αυτά είναι σημαντικά και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, αυτό είναι πάλι άλλου είδους θέμα, άλλου παπά Ευαγγέλιο. Ο κύριος Βανόρντεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλουμε τίποτα να υποβαθμίζω τη συζήτησή μας που είναι πάρα πολύ σοβαρή γιατί ε, βασικά γκρινιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχει ως θεμέλιο ένα αφήγημα αναλυθές και ότι δηλαδή αυτό κάνει, κάνει προπαγάνδα εις βάρος του λαού. Και λένε ότι για όλα τα προβλήματα η Πανάκια είναι περισσότερη Ευρώπη. Αλλά όταν βλέπει λοιπόν κανείς αυτό το θέμα που τώρα συζητούμε από πλευράς Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει κανεί να καταλάβει πώς είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι θα έπρεπε να κάνει. Άρα θα πρέπει να δούμε ε, τι γίνεται με τις ελευθερίες, ε, την πραγματικότητα της κοινωνία μας, γιατί τελικά ε, εντάξει, δεν, τίποτα δεν είναι νέο. Αυτά τα γνωρίζουμε και ξέρουμε πώς λειτουργεί η, Σοβιετική, η ρωσική ψυχή και πριν από τη Σοβιετική Ένωση. Ξέρουμε ποιος είναι ο κύκλος της ζωής στην ε, Σοβιετική Ένωση ή στην Ρωσία. Και επίσης ε, συμφωνώ με αυτό το οποίο ελέγχθη από τον κύριο Πάσχο για ε, το που είμαστε ευάλωτοι, η Ρουμανία πούμε, και η Βουλγαρία που είναι τελικά οι γείτονες της ε, Ρωσίας. Στο think tank που συμμετέχω έχουμε εκπονήσει και δημοσιεύουμε μια μελέτη για την Βουλγαρία που ακριβώς θίγει αυτά τα οποία σήμερα συζητούμε ότι θα πρέπει δηλαδή να προσέξουμε περισσότερο εκείνες τις ε, χώρες που είναι οι πιο ευάλωτες όσον αφορά αυτή την συνεχή ομοβροντία ρωσικής προπαγάνδας. Επίσης, συμφωνώ με αυτό το οποίο τονίσατε ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερο συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών ε, υπηρεσιών και φορέων. Συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να κάνει ε, αυτά τα οποία θα έπρεπε να γίνονται αλλού ή γίνονται αλλού όπως ας πούμε στο ΝΑΤΟ. Άρα θα πρέπει να κάτσουμε και να σκεφτούμε καλά ποια θα πρέπει να είναι η κατανομή των αρμοδιοτήτων. Επίσης, και αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ λεπτό και δύσκολο, να δούμε πώς θα ελκύσουμε την προσοχή της ρωσικής κοινή γνώμης. Ίσως θα πρέπει να βρούμε κάποιο κοινό παρονομαστή, κάποιο κοινό τόπο, ίσως ας πούμε αυτό εκπλήσει σε πρώτη φάση, αλλά ας πούμε να, η τρομοκρατία η Ισλαμική. Αυτό είναι κοινό ενδιαφέρον ή συμφέρον της δύση και ε, της ε, Ρωσίας. Άρα εκεί θα πρέπει να πατήσουμε και να το εκμεταλλευτούμε περισσότερο. Ευχαριστώ τους μιλητές, αλλά θα πρέπει και εγώ να φύγω γιατί θα πρέπει να προεδρεύσω στην ε, συνεδρίαση της αντιπροσωπείας μας για τις σχέσεις με την Ινδία. Πρέπει να έχουμε αρχίσει εδώ και ένα δεκάλεπτο. Σας ευχαριστώ λοιπόν, Κούζα. Κατά τη γνώμη μου, ξέρετε, θεωρώ ότι πρόκειται για οπισθοδρόμηση. Μιλάμε για μακαρθισμό, μιλάμε για ψυχρό πόλεμο. Όταν μιλάμε για τα ΜΜΕ και έχουμε τέτοιου είδους αντιπαράθεση, τότε δαιμονοποιούμε τα μέσα ενημέρωσης και στοχοποιούμε τους δημοσιογράφους πάντω, αντί να ανησυχούμε για την συγκέντρωση των ΜΜΕ, ε, θα έπρεπε να ψάχνουμε αντίβαρα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε εγγυήσει πλουραλισμού. Να δούμε τι γίνεται με τις συνθήκες εργασίας των ε, δημοσιογράφων. Υπάρχουν τόσες καταγγελίε. Αυτό έπρεπε να δούμε σαν Ευρωπαίοι. Μην ε, γελιόμαστε. Εδώ πρόκειται για πόλεμο πληροφορίας. και ξέρουμε ότι εάν χαθεί ο έλεγχος τη πληροφορία είναι σαν να χάνεται ένας πόλεμος. Είδαμε τι έγινε και με την Βρετανία. Να και στον πόλεμο του ε, κόλπου. Το, είχαμε μόνο το CNN. Δεν υπήρχαν δημοσιογράφοι εκεί επιτόπου να, να γράφουν και το CNN. Επομένως, ε, ξέρουμε τι έκανε. Ήταν μία μόνο φωνή που έκανε προπαγάνδα. Το ίδιο και στην Ιουγκοσλαβία. Είχαμε 16 δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν όταν έγιναν οι βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ στο Βελιγράδι. Και ε, επίσης αποφάσισε το ΝΑΤΟ επίσης ε, ε, ποιοι είναι οι κακοί και ποιοι οι καλοί δημοσιογράφοι. Το ίδιο και στο Αφγανιστάν. Και εκεί είχαμε CNN και βομβαρδισμούς κατά τον ΜΜΕ στην Καμπούλ. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι σαν να έχουμε μια τρίμπιουν, μια χέρα τρίμπιουν ευρωπαϊκή. Το ίδιο έγινε και ε, στο Αφγανιστάν, το ίδιο έγινε και αλλού με τους ε, πεζοναύτες. Αυτό το οποίο κάνουν δεν υπήρχε πόλεμος, οπότε ε, είχαν ε, ε, επιτεθεί στα ΜΜΕ, ας πούμε στο Αμπουντάμπι, στο Reuters, τρεις δημοσιογράφοι. Αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρχουν περισσότεροι εξάρτητοι δημοσιογράφοι και δημοσιογραφία και λιγότερες δολοφονίες. 400 δημοσιογράφους που έχουμε ε, μέχρι τώρα νεκρούς, δηλαδή ένα ρεκόρ. Και ε, αν δεν ήταν το CNN θα, θα ήταν το, το, το UPC ή θα είναι το Russia Today. Και εγώ δεν, σα σας τα λέω. δεν σας τα λέω σαν ε, ε, ευρωβουλευτής μόνο. Θα πρέπει να πούμε ποιος είναι ρωσόφοβος και ποιος είναι ε, φίλος της Ρωσίας. Δεν είμαστε χαζοί, δεν έχουμε ανάγκη που κάνουμε μεγάλο αδελφό να μας πείτε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Στάτινα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί, προσκεκλημένοι μας. Είναι πολύ θετικό το ότι εδώ και μας τα είπατε. Εσείς είστε μοναχικοί οδηπόροι και μαχητές σε αυτόν τον πόλεμο της πληροφορίας. Πρόκειται για μία μάχη άνηση. Και θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι. Τον κύριο Πόρτμαν. Το επιτελείο σας έχει ως αφετηρία την εντολή της κυρίας Μαγκερίνη ή κάποιο άλλο ενωσιακή πρωτοβουλία ή κάποιο πρωτοβουλία του Συμβουλίου, έτσι δεν είναι. Α, από ό,τι κατάλαβα έχετε εννέα άτομα στην ομάδα σας. Όμως, για να καθίσετε και σκεφτείτε τι διαθέτει η Ρωσία. Είναι πάρα πολύ άνηση η μάχη, δεν έχετε αρκετούς ε, πόρους. Θα πρέπει ομένως να μην υποτιμούμε το πόσο σημαντική είναι η δουλειά σας στο να φρενάρετε ε, αυτές τις ε, προσπάθειες παραπληροφόρησης, αυτόν τον πόλεμο της πληροφορία. Θα πρέπει επομένω καλύτερα να λειτουργεί η προσπάθειά μας κατά της ε, προπαγάνδα. Ό,τι για πέστε μας, πώς γίνεται η χρηματοδότησή σας, έχετε κράτη-μέλη που ορίζονται από τα ε, κάποια, κάποια μέλη στην ομάδα που γυρίζονται από τα κράτη-μέλη τι, τι έχει να σα στηρίξει σε αυτή τη μοναχική σας πορεία Πρόεδρο Φροντζούλικα Κυρίες και κύριοι μιλούμε για παραπληροφόρηση και για αυτόν τον πόλεμο πληροφορία αυτόν τον βρώμικο πόλεμο που έχει κηρύξει η Ρωσία Έχετε ακούσει την στρατιωτική επανάσταση στην Ρωσία που ξεκίνησε το 2008 μετά τα επεισόδια με την Γεωργία. Αυτό θα ολοκληρωθεί το 2020 και έχουν γίνει πάρα πολλές εξελίξεις τώρα όσον αφορά νέα όπλα και τεχνολογία. Ε, αυτός ο χρονικός πόλεμος είναι τμήμα αυτής της στρατιωτικής επανάστασης της Ρωσίας. Ξέρετε, την πρώτη μέρα που άρχισε ο πόλεμος με την ε, Γεωργία είχαμε κατάρρευση τριών αεροπλάνων και άλλων τεσσάρων την επόμενη μέρα. Είχαμε ακόμα και φίλια πειρά Αλλά βέβαια τελικά κατατρόπωσαν οι Ρώσοι τους Γεωργιανούς. Πρόκειται για αυτή την επανάσταση η οποία θα πρέπει να αναχαιριστεί. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε πως η Δύση και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να φρενάρει αυτή την Ρωσική Επανάσταση. Τι γίνεται με τα δυτικά κόμματα. Επιδοτούνται, όπως επιδοτούνται και κάποιες οργανώσεις, κάποια μέσα ενημέρωση από τη Ρωσία. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε τρεις πολύ σημαντικές χώρες που εάν πέσουν τότε θα έχουμε μια καταστροφή για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδίω την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλώ για Ουκρανία, Μολδαβία και Γεωργία. Και στις τρεις αυτές χώρες η Ρωσία ενισχύει πολιτικούς και πολιτικά κόμματα. Κάνουν ό,τι μπορούν για να υπονομεύσουν το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε αυτές τις ε, χώρες, τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα τους πολιτικούς, τους φιλοευρωπαίους οργανισμούς, μέσα ενημέρωσης θέλω να σας πω μόνο το εξής είναι σημαντικό να εξηγείτε στον κόσμο το τι κάνει η Ρωσία αλλά ταυτόχρονα κυρίες και κύριοι να μην ξεχνούμε τον κόσμο στη Ρωσία να μην μπερδεύουμε την ρώσικη κυβέρνηση με το ρωσικό λαό ο λαός θα πρέπει να καταλάβει και αυτό είναι δουλειά των δικών σας φορέων, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι εναντίον τους να καταλάβουν ότι οι καλύτερες σχέσεις Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι προς το συμφέρον τους για μια καλύτερη ζωή που θα είχαν εάν η Ρωσία είχε καλύτερες σχέσεις με Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα πρέπει να εξηγηθεί στους Ρώσους πολίτες και αυτό είναι δική σας αποστολή και όχι η προπαγάνδα γιατί το 1880 είπαν στο Γεύσκι περίπου ότι εμείς οι Ρώσοι σας θεωρούμε σαν του Μογγόλους αλλά εμείς εδώ στην Ασία είμαστε οι πραγματικοί Ευρωπαίοι θα πρέπει ομένως να εξηγηθεί στου Ρώσους ότι μόνο η συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ένωση θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι προ το συμφέρον του. Ο κύριος ε, Μαρακιουρικέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις ε, πληροφορίες που μας ε, δώσατε και για τη δουλειά που κάνατε. Η δουλειά που ξεκινήσατε πρέπει να επεκταθεί. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η Ρωσία προσπαθεί να επιτεθεί στα μέσα της Δύσης και εμείς δεν κάνουμε τίποτα για να αποδομήσουμε την ρωσική προπαγάνδα να την αποδομήσουμε ε, κυρίως εκείνη που απευθύνεται προς τη Δύση ε, που έχει ως στόχο να ε, προβάλλει το καθεστώς του Πούτιν. Η Ρωσία λέει ότι συνεχίζει τον αγώνα κατά του φασισμού αυτό 70 χρόνια μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και λέει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν αντικομουνιστικές δυνάμεις αλλά όλα αυτά δεν είναι αλήθεια ε, η αλήθεια είναι ότι το καθεστώς της Ρωσίας είναι ένα μετακομμουνιστικό καθεστώς το δόγμα του στρατηγού Γκρασίμοφ είναι τα γνωστά αναθερμένη την ρωσική ε, προπαγάνδα ε, μεταθέτει το ενδιαφέρον από αυτά που κάνουν οι Ρώσοι στα ανθρωπιστικά προβλήματα. Αυτή κατ' ουσίαν ήταν και η ρωσική προπαγάνδα κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ. Δηλαδή εστίασαν εκεί ε, στις αποτυχίες της δύση. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε πάλι την ίδια προπαγάνδα ενώ ε, υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα. Υπάρχει άλλο πρόβλημα, το μεταναστευτικό. Ε, προσπαθούν λοιπόν να μεταθέσουν την προσοχή των πολιτών από τα ουσιαστικά προβλήματα. Η δική μας λοιπόν ευθύνη ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Και ας μην ξεχνάμε ότι στην Ουκρανία ή και στη Γεωργία μένεται πόλεμος ε, για να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία αυτών των κρατών. Καταρχήν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση. Κυρίες και κύριοι, εφόσον εμφανίζονται τέτοιου είδους προβλήματα εφόσον υπάρχει πρόταση ψηφίσματος πρέπει να επισημάνουμε ότι οι Μπολσεβίκοι αντιμετωπίζονται, αποθεώνονται στη Ρωσία, ενώ τα περισσότερα μέλη εδώ του Κοινοβουλίου δεν αποθεώνουν τη ρωσική ιστορία, κάθε άλλο. Τα χέρια μας όμως είναι δεμένα. Γι' αυτό λοιπόν είτε θα πρέπει να αποδείξουμε ποιες είναι οι προσπάθειες ε, του Πούτιν ή θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι υπάρχει ε, μια ολιγαρχική δομή που είναι σαν να λέμε άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Αν λοιπόν ε, δεν το επισημάνουμε αυτό. Δεν επισημάνουμε ότι στη ε, Ρωσία υπάρχει ένας νέος ε, πολιτισμός όπου αποθεώνονται οι ολιγάρχες. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον παλαιό πολιτισμό. Αν δεν τα επισημάνουμε όλα αυτά, δεν επισημάνουμε τις ανθρωπιστικές αξίες, τότε δεν θα τα καταφέρουμε. Κυρία Νικολάη. Εντάξει, μπορεί να είμαι και κύριος μερικές φορές. Λοιπόν, να συγχαρώ ε, για τη συζήτηση που είναι πολύ επίκαιρη. Δεν είναι κάτι αφηρημένο. Δεν μιλάμε για το μέλλον, εδώ μιλάμε για την πραγματικότητα. Και για τις τέως κομμουνιστικές χώρες. Και ε, κάποιες φορές ε, νιώθω σαν να είμαστε στόχος αυτής της προπαγάνδας. Είναι τεράστιο πρόβλημα για μας. Γιατί κάποιες φορές δεν ξέρουμε. Ο κύριος ε, Γερασίμοφ είναι ο Γκάιτιν. Ποιος, ποιος βρίσκεται πίσω από αυτή την προπαγάνδα. Αν οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι έχουν αυτή την προσέγγιση, για αυτό το λέμε ένα συμμετρικό πόλεμο, Πρέπει και εμείς εδώ στην Ευρώπη να προστατεύσουμε τις ε, αξίες μας. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα μέσα ενημέρωσης και επιτρέπουμε την ελευθερία της έκφρασης και του λόγου, άρθρο 2 της συνθήκης, αλλά πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εμείς στην Ευρώπη αυτό το πρόβλημα. Δεύτερο ερώτημα, στο τέφαρ θαλασσιοδόγμα, όπως αναθεωρήθηκε τον Ιούλιο του 2015 από τη Ρωσία. Γνωρίζουμε όλοι ότι έχουν κάποιες ζώνες ε, όπου δεν υπάρχει τα πρόσβαση, ε, στη Βόρεια Θάλασσα κυριαρχούν. Και αν δούμε τι γίνεται με Ρωσία, Τουρκία, απόφαση ΝΑΤΟ κτλ, Το διεθνές δίκαιο, πώς το βλέπετε, έχουμε τη σήμαση Μοντρέ, που είναι πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά ξένα, ξένες δυνάμεις να εισέρχονται στα χωρικά της Βόρειας Θάλασσας, στη Βόρεια Θάλασσα. Επιτρέψτε μου ευθύς εξ αρχής μια Λοιπόν, ε, επιτρέψτε μου να προτάξω το εξής. Ε, κοιτάξτε, εγώ τη ε, ρωσική πολιτική την αντιμετωπίζω κάπως διαφοροποιημένο από ό,τι όλοι οι άλλοι. Δηλαδή, το τι σχέση έχει η σημερινή Ρωσία με τον κομμουνισμό το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Και όσον αφορά την τρέχουσα πολιτική της Ρωσίας και τις σχέσεις της με τις ακραίες τάσεις και αυτό το γνωρίζω και σε πολλές περιπτώσεις το επικρίνω. Δεν αμφισβητώ αυτά που ελέγχθησαν, όμως ε, θέλω να σας επισημάνω κάτι που έχει λεχτεί η αλήθεια που ελέγχθη ότι η αλήθεια είναι το πρώτο θύμα του πολέμου. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Θα έπρεπε να είναι η πρόταση, η αλήθεια είναι το πρώτο θύμα πριν από το ξέσπασμα ενός πολέμου και είναι και το πρώτο θύμα σε όλες ε, τις συγκρουσιακές καταστάσεις. Άρα δηλαδή ε, όλα αυτά το βρίσκω παράλογο να τα ανάγουμε μόνο στη Ρωσία. Ε, αναλύσεις που ακούστηκαν είναι χρήσιμες, αλλά θα με ενδιαφέρει παραδείγματο χάρη και μια ανάλυση που να αφορά τη Γερμανία για την εικόνα εχθρού που συσχετίζεται με τη Ρωσία. Και δεν είναι αυτό κάτι καινούριο, ότι δηλαδή μυστικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο κάνουν προπαγάνδα και αυτό είναι ένα σκέλος ε, ενός πολέμου. Και γι' αυτό λοιπόν ε, κάποιες ε, ομότητες και βιότητες που διαπράχτησαν στην, στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας αποδείχτηκε ότι ήταν ψέματα ή αν θέλετε τα όπλα μαζικής ε, καταστροφής του Σαντάμ Χωσήν αποδείχτηκε ότι ήταν ψέμα αλλά μετά πια εκ των υστέρων ε, σκασίλα τους όλοι δεν τους ενδιέφερε ε, ήταν όλα αυτά μέσα στο παιχνίδι και εκ των υστέρων κανείς δεν ενδιαφερόταν έχω κάνει και εγώ τη δική μου την προσωπική εμπειρία ας πούμε στη γερμανική τηλεόραση έχω δώσει συνεντεύξεις για την περίπλοκη κατάσταση στην Αρκτική. Ξέρουμε πόσο περίπλοκη είναι εκεί η κατάσταση, ε, πώς ε, υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα, οικολογικά, οικονομικά συμφέροντα. Αυτή η συνέντευξη, ξέρετε τι τίτλο είχε εκ των υστέρων, «Ο φόβος της Βόρειας Ευρώπης από τη Ρωσία ή σε σχέση με τη Ρωσία και ό,τι εγώ προσπάθησα να πω για να δείξω πόσο περίπλοκη ε, είναι η κατάσταση αυτά είχαν εξαφανιστεί. Βεβαίω αυτό που σας λέω ήταν πολύ πιο υφέρπον σε υφέρπουσα μορφή από αυτά που ακούσαμε αλλά εν πάση περιπτώσει να το δεχτούμε και αυτό ότι υπάρχει και η δυτική προπαγάνδα. Κύριε Γκάλερ, εγώ δεν τα εξισώνω, δεν τα ισοπεδώνω όλα. Λέει πρόεδρο, εντάξει, τώρα μην κάνετε και διάλογο. Εγώ απλά Λέω τη γνώμη μου γιατί για μένα είναι σημαντική. Δεν τα βάζω όλα στο ίδιο καζάνι, αλλά κύριε Γκάλερ, εγώ λέω το εξής, ότι δεν πρέπει ε, να είμαστε κομμάτι του μηχανισμού προπαγάνδας. Και το είπατε κι εσείς και εγώ, δεν θέλω να βρούμε ε, άλλα μέσα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι λάθος. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αγωνιστούμε έτσι ώστε οι δημοσιογράφοι σε ολόκληρο τον κόσμο να έχουν σωστές συνθήκες εργασίας, να έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν την αλήθεια. Και αυτό που είπατε εσύ δεν το βρίσκω σωστό, που είπατε ότι οι άνθρωποι ε, βρίσκουν ε, ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν να ε, επιβεβαιώνονται σε αυτό που ήδη πιστεύουν. Άρα δηλαδή εγώ καταλήγω στο ότι όλα αυτά οδηγούν σε πόλωση και δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος ε, όπου δηλαδή τώρα εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε ότι και εμείς ε, πρέπει να έχουμε μια προπαγανδιστική, προπαγανδιστική μηχανή που να τη χρησιμοποιούμε οποτεδήποτε αυτή είναι απαραίτητη. Ο κύριος Φρόιντ, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις. Βρίσκομαι σε κάπως δύσκολη θέση γιατί διατέλεσα δημοσιογράφος στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου και έγινα πολιτικός ε, μόλις ε, στις αρχές του 2014. Δεν θέλω λοιπόν σε καμία περίπτωση να υπερασπιστώ αυτό που λέτε για τη ρωσική προπαγάνδα, ούτε να δημιουργήσω κάποια αντιπαράθεση. Αλλά θα αντιπαραβάλλουμε αυτό με το πολύπλοκο περιβάλλον το επικοινωνιακό εδώ, στη Δύση. Αν δούμε τα τελευταία δημοσιεύματα για τους πρόσφυγες, Και πρέπει να πω ότι σε πολλά μίντια ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά ε, λάθη και ψέματα. Αυστριακός τύπος για παράδειγμα που κατηγορεί ότι οι πρόσφυγες καταστρέφουν τις ταλέτες στα τρένα, μα δεν έγινε ποτέ αυτό. Ότι κλέβουν από σούπερ μάρκετ, ούτε και αυτό έχει γίνει ποτέ. Αν όμως το γράψει μια εφημερίδα, το αναπαράγουν και επόμενες, υπόλοιπες. και πολλές φορές, ε, ακόμη και αν δεν υπάρχει βάση για κάποιο δημοσίευμα, το ένα εντυπώ αναφέρεται στο άλλο, ως πηγή. Μέχρι και μένα με κατηγόρησαν το ε, τελευταία ε, εβδομάδα της προεκλογικής εκστρατείας ότι ήμουν κατάσκοπος και αυτό το αναπαρήγαγαν όλες οι αυστριακές εφημερίδες ότι ήμουν κατάσκοπη για την πρώην Κοσλαβία Στην πρώην Κοσλαβία τέλος πάντων. Και τελικά όχι δεν ήμουν εγώ κατάσκοπος, αλλά εμένα με κατασκοπεύανε. Αυτό αποδείχτηκε. Τέλος πάντων, έτσι, η Ρίστο, είναι παρόδο. Αυτό ε, πώς πέρασε όμως ε, στον τύπο, ε, δύο γραμμούλες κάπου σε ένα μικρό αρθράκι για την κυρία Λέζιν που μίλησε για τα όπλα μαζικής καταστροφής που ο Κόλιν Πάουελ είχε παρουσιάσει ε, στα Ηνωμένα Έθνη. Όμως πήραν την ιστορία και τα μέσα ενημέρωσης και δεν είπαν ότι οι μεγάλες δυνάμεις, ε, όχι μόνο ο Κόλιν Πάουλ αλλά και ο αντιπρόεδρος Ντικ και όλοι οι άλλοι που είχαν πολύ στενές σχέσεις με τα μέσα, ότι αυτοί έδωσαν αυτή την, την ιστορία και τη φούσκωσαν. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν ασκούμε κριτική σε άλλες χώρες και στον τύπο ε, άλλων χωρών. Πρέπει να δούμε τι κάνουν και τα δικά μας μίντια. Και αυτά θα μπορούσαν να δεχθούν άνετα κριτική. Τέλο πάντων, ε, υπάρχουν και άλλα δύο-τρία πράγματα, αλλά να μην μακρηγορήσω άλλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Ευχαριστώ, κύριο Μποστινάρου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ την Πρόεδρο για τη διοργάνωση αυτή τη πολύ σημαντική συνάντηση. Είναι επίκαιρη, αλλά όχι ακριβώς επίκαιρη, γιατί όλο και καινούριε εξελίξεις έχουμε και Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε. Η δύναμη, η δυνατότητα και η βούλησή μας φαίνεται να είναι και αδύναμη και να μετριάζεται όλο και περισσότερο. Τέλος πάντων, να σας πω κάτι που όλοι το γνωρίζουμε, την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι θα δημιουργηθεί μια δυνατότητα για την αντιμετώπιση της ρωσικής προπαγάνδας. Ε, αυτή ήταν μια μεγάλη υπόσχεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν ακολουθήθηκε όμως ε, από κάτι συγκεκριμένο. Μέχρι τώρα δηλαδή πολύ απλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αντιμετώπισης της ρωσικής προπαγάνδας. Από την άλλη πλευρά όμως ταυτόχρονα και εδώ θέλω να αναφερθώ σε κάτι το οποίο ε, γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο που στο Channel One κατηγορήθηκαν ότι διαστρεβλώνουν και προωθούν ε, ψευδείς ε, πληροφορίες και κάνουν προπαγάνδα. Έγινε μια, ε, υπήρξε μια απόφαση και την γνωστοποίηση στο Κογκρέσο και ο αρχηγός της CIA ότι πρέπει να ερευνηθεί η χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων στην Ευρώπη από τη Ρωσία, που στόχο έχει να διαιρέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπονομεύει τις σχέσεις της Ένωσης με τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ. Αν αυτό ανακοινώθηκε στο Κογκρέσο, με τον κύριο Κλάπερ να είναι ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και αν συζητηθεί και στο Κογκρέσο αυτή η έκθεση και ακολουθήσουν και κάποιες συγκεκριμένες δράσεις, μπορεί η Ευρώπη να είμαστε τόσο εδώ ήρεμοι, χαλαροί, να μην βλέπουμε τι συμβαίνει και να μην κάνουμε κάτι για να προστατευτούμε, να εξασφαλίσουμε κάποιο είδους ασυλία, διότι δεν βλέπω να υπάρχει κάτι τέτοιο. Η Ευρώπη, Ευρώπη ΝΑΤΟ, μπορούν από κοινού να κάνουν κάτι για να αντιμετωπίσουν την προπαγάνδα και τη ρωσική πολιτικών κομμάτων. Πριν δύο-τρει μέρε διάβασα ότι ο Γενικό Αγγελέα ε, στη Γερμανία ερευνά αφενός χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από την ακροδεξιά και την ακροαριστερά. Και φυσικά γιατί δεν θέλω να αφισβητήσω την προσήλωση και τη συλλογιστική βάση της οποίας ο Γενικός Αγγελάς το αποφάσισε. Αλλά βλέπουμε αυτό από τη μία και από την άλλη τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η ΜΚΟ και η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων αντιμετωπίσετε από τη Ρωσία ως κομμάτι αυτού του βρεδικού πολέμου. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ούτε έγινε κατά λάθο. Είναι τμήμα μιας ολόκληρης στρατηγικής. Καταλαβαίνω ότι η Ρωσία κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Αλλά δεν καταλαβαίνω εμείς τι κάνουμε. Εμείς στη Δύση, εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δείχνουμε τέτοια προθυμία να προστατευτούμε, να δημιουργήσουμε μια δυνατότητα και μια δομή που θα μας προστατεύει. Υπάρχει και αυτή η προσπάθεια διέρεσης. Υπήρξε αυτή η υπόθεση στη Γερμανία με ένα κορίτσι δεκατεριών ετών και ένας βουλευτής στην Bundestag, διακεκριμένος βουλευτής, είπε ότι ο στόχος ήταν η αποδυνάμωση της θέσης της Γερμανίας Καγκελαρίου. Άρα να αποδυναμωθεί η Ευρώπη να δράσει. Αυτός είναι ο τελικός στόχος. Δεν είμαι Γερμανός εγώ, αλλά δεν θα διστάσω να πω ότι είναι σημαντικό αυτό. Και αν θεωρεί ότι έτσι έχουν τα πράγματα η Bundestag, η Ευρώπη τι πρέπει να κάνει. Να μείνει σε αυτή την επικίνδυνη αδράνεια ε, και νυφαλιότητα και χαλαρότητα και να μην αντιμετωπίσει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επιβλαβές για την ίδια την επιβίωση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Πρέπει και εμείς από την πλευρά μας να δημιουργήσουμε τις δυνατότητες και τις δομές για να αντιμετωπίσουν αυτή την πραγματικότητα που είναι ένα κομμάτι του υβριδικού πολέμου που στόχο έχει να μας διαρρέσει, να μας αποδυναμώσει και γιατί όχι να προετοιμάσει και την ίδια την κατάρρευση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Αν αυτό δεν το καταλάβουμε, τότε αξίζει να δούμε και την άλλη όψη τη πραγματικότητα μετά. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αυτή είναι η πραγματικότητα και απαιτεί δράση. Mr. Indrek Tarand, then myself, and the list is closed. Ο επόμενο ομιλητή. Και κατόπιν θα μιλήσει υποφαινόμενη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάντοτε η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ξέρετε κατά πολλούς τρόπους μπορεί κανείς να ε, δώσει τον ορισμό της ε, παρερμηνίας, των ε, μικρών μεγάλων ψεμάτων, της παραπληροφόρησης, της προπαγάνδας κλπ. κλπ. Όμως εγώ θα ήθελα θα ήθελα να προσθέσω μια πινελιά αισιόδοξη σε αυτή τη ε, συζήτηση. Για ακούστε προσεκτικά. Εγώ 27 χρόνια ζω με την ρωσική προπαγάνδα. Ακόμα όμω το μυαλό μου, το μισό μυαλό, μισό εγκεφαλός μου ακόμα λειτουργεί. Και ξέρετε ήδη στο σχολείο ε, όλα αυτά ε, γίνανε. Είχαμε έναν επίσκοπο από το Νόβγκοροντ ο οποίο πήγε στην Ιερουσαλήμ, ξαναγύρισε, ήταν Ρώσος. Τέτοιος είχαμε και ε, το χειριστήκαμε ως εξή. Δεν προσπάθησαμε να ανταγωνιστούμε ε, τα κομμουνιστικά ΜΜΕ, ούτε φωνάξαμε τη, τη Δύση. Το αντιμετωπίσαμε με χιούμορ και θεωρώ ότι αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο επιβίωση. Α, οπότε... Να, τελικά θα πρέπει κανείς να βάλει τα γέλια για τις προσπάθειες του Πούτιν να κάνει πλήση εγκεφάλου στην Ουκρανία, τη Γεωργία κλπ. Άρα, τελικά αυτοί έχουν το πρόβλημα. Αυτοί δεν μπορούν να έχουν σωστή πληροφόρηση. Εμεί έχουμε πολλέ πηγέ πληροφόρηση. Αν θέλουν να κάνουν την κοινωνία του σαν τη δική μα, θα του βοηθήσουμε. Αν θεωρούν ότι θέλουν ε, διαφθορά και αν νομίζουν ότι η δημοκρατία και η μεταρρύθμιση πρέπει να πει κανεί να βάλει στη φυλακή του μεταρρυθμιστέ όπω γίνεται στη Γεωργία, ε, τι να κάνουμε τότε. Ε, δικαίωμά του είναι να κάνουν τι επιλογέ του. Ευχαριστώ. Η πρόεδρο, σα ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσω και εγώ και του τρει εμπειρογνώμονες για το εξαιρετικό του ε, έργο και τις εισηγήσεις τους. Μπράβο, ήταν πάρα πολύ ενημερωτικά όλα αυτά, ε, ήταν πάρα πολύ ακριβή και νομίζω ότι πρόκειται για μια μεθοδολογία κρυστάλλινη όσον αφορά του τι γίνεται από την Stratcom, τι γίνεται με την ρωσική δράση, με την προπαγάνδα για την περίοδο πριν την εισβολή στην Ουκρανία. Τι έγινε κατά την εισβολή, αλλά και το τι έγινε μετά <clears throat> κατόπιν της ε, προσάρτησης της Κρυμαίας. Εμείς δεν θέλουμε να επικρίνουμε τα μεσενημέρωσης. Τα μεσενημέρωσης χειραγωγούνται, χρησιμοποιούνται. Και ξέρουμε τι γίνεται με τα μεσημέρωση, όχι μόνο στη Ρωσία αλλά και στι δικές μας χώρες. Και δεν πρόκειται μόνο για Βουλγαρία, Πολωνία, Βουλγαρία. Αλλά σε πάρα πολλές χώρες έχουμε τέτοια φαινόμενα και σε πολλές χώρες του ΝΑΤΟ. Οπότε και έχουμε τέτοια εργαλεία, εργαλεία επιρροής της κοινωνίας μας. Έτσι βλέπω εγώ τα πράγματα. Και βασικός στόχος τους είναι να διασπάσουν την ενότητά μας. Και χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ όπως χρησιμοποιούν και την ε, χρηματοδότηση κάποιων κομμάτων. Αλλά έχουμε ένα σωρό πολιτικούς που είναι σε πολλά κόμματα και οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια τα παίρνουν από τους Ρώσους. Εδώ και χρόνια δεν τα ξέρουμε αυτά. Πρόκειται για ε, παλιούς, δοκιμασμένους, έμπειρους πολιτικούς. Γνωστά είναι όλα αυτά. Δεν θα πρέπει να βρεθεί ένα τρόπο να το ανασχέσουμε αυτό, γιατί ένα από του μύθου αυτή τη ε, στατική επικοινωνία των Ρώσων είναι το εξή. Αυτό ο μύθο τη ε, ρωσική υπερδύναμη, οικονομική και στρατιωτικής. Και σε τέτοια εποχή επιθετικότητας, ε, παρέμβασης, εμπλοκής όπως και να το πείτε για την Ουκρανία. Είναι ξεκάθαρα περίπτωση επιθετικότητας. Αλλού προσπαθούν να δημιουργήσουν μια πολύ θετικότερη εικόνα. Επίσης θα πρέπει να δείξουμε στην κοινή γνώμη της δική μας αυτό το οποίο θέλω να πούνε δηλαδή η ρωσική αγορά είναι η πιο μεγάλη και η πιο πλούσια για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αυτό είναι πρόβλημα γιατί κάθε φορά θα πρέπει εμείς να μπορούμε να αντιδράσουμε με στοχευμένο τρόπο. Είναι δύσκολη η οικονομική συγκυρία. Ε, αλλά θα, θα πρέπει να πούμε ότι η ρωσική οικονομία μπορεί να, πρέπει να συγκριθεί με την οικονομία των κάτω χωρών, τίποτε παραπάνω. Και είδαμε το πόσο ισχυρή είναι η στρατηγική μηχανή της Ρωσίας στον πόλεμο με την Γεωργία. Καλά, καλά, βελτιώθηκε, αλλά όχι και πάρα πολύ. Επίσης, είναι και το θέμα των αποδειχθούν οι σχέσεις Σοβιετική Ένωσης και της σημερινής Ρωσία γιατί είναι από του μύθους τη πολιτικής του Πούτιν. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Να συνδέσει την Ρωσία του με την Σταλινική Σοβιετική Ένωση. χρησιμοποίησε τα σύμβολα του σταλινισμού το 2010 τότε που είχε τον εορτασμό για την νίκη κατά του χιτλερισμού. Αυτό ήταν δύσκολη στιγμή για την Πολωνία. Γιατί ακόμα, ακόμα να ανακαλύπτουμε τάφους εξεχόντων Πολωνών που δολοφονήθηκαν από τους Σοβιετικούς. Επομένως, εκεί είναι το πρόβλημα το πόσο προσπαθεί να οριοποιήσει ο Πούτιν ε, την σταλινική κληρονομιά. Και τώρα με την ίδια σειρά που έκανε τις του να έχουν το λόγο οι καλεσμένοι μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που είπατε. Θα μου επιτρέψετε να επανέλθω σε ορισμένα θέματα. Έχουν γίνει διάφορες παρεμβάσεις όπου έγινε λόγος για το ότι είναι απαραίτητο ε, να αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία στην κοινή γνώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε, αναπτύσσοντας το δίκτυό μας ε, εκείνων που έρχονται σε εμά και μας ενημερώνουν για την παραπληροφόρηση. Σας λέω, ε, υπάρχει βέβαια και ένα όριο ως προς το πόσο μπορεί η υπηρεσία εξωτερικής δράσης να διεισδύσει στους πολίτες χωρίς τη βοήθεια των κρατών μελών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τη δική σας τη βοηθεία να στηρίξετε το δίκτυό μας και να ε, διαδώσουμε σωστά τις πληροφορίες. Υπάρχουν και κάποια άλλοι στόχοι έχουμε ε, τους ανθρώπους μας στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης και ε, κυρίως ε, Ουκρανία, Γεωργία, Μολδαβία. Αλλά εστιάζουμε την προσοχή μας και σε άλλες χώρες και φτάνουμε μέχρι και την Κεντρική Ασία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Όπως σας είπα όμως θέλουμε να απευθυνθούμε σε ρωσόφωνους εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε τέτοιο ένα ερώτημα ε, μήπως υπάρχει επικάλυψη ε, προσπαθειών, μήπως θα πρέπει να υπάρχει καλύτερο συντονισμό Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι εδώ υπάρχει ένα κενό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν ε, ανταποκνόταν, αλλά όσον αφορά το συντονισμό, συντονιζόμαστε πολύ στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και με το ΝΑΤΟ, γιατί ε, οργανώνουμε από κοινού ασκήσεις, ανταλλάσσουμε πληροφορίες, προϊόντα, τα διάφορα προγράμματα τα κάνουμε από κοινού και έτσι ο ένας επωφελείται από τον άλλον. Και τέλος, ε, ο κύριος Στετίνα ε, υπέβαλε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Να απαντήσω λοιπόν πράγματι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαρτίου του περασμένου έτους ε, οδήγησαν την ύπατη εκπρόσωπο να καταρτήσει να συστήσει αυτή την ομάδα. Εννέα άνθρωποι είμαστε, όπως σας είπα. Δεν προκαλούμε κόστος, δεν έχουμε επιπρόσθετο προϋπολογισμό και δεν έχουμε επιπρόσθετο προσωπικό. Δηλαδή ε, χρησιμοποιούμε το προσωπικό ε, που ήδη υπήρχε, έναν από την Κομισιόν, ένα από το Κοινοβούλιο και έχουμε πέντε κράτη-μέλη, Βασίλειο, Δανία, Τσεχία, Λετωνία και Εστονία που μας στηρίζουν. Έχουμε πολύ μικρά ποσά από τον προπλογισμό Stratcom της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ε, εποφελούμεθα βέβαια από την Κομισιόν 11 εκατομμύριο ευρώ είναι ο προπολογισμός της ε, για την, σχέση, την εταιρική σχέση με τις ανατολικές χώρες. Εν πάση περιπτώσει εμείς όπως σας είπα είμαστε μια μικρή ομάδα που δεν επιβαρύνει οικονομικά. Ο κύριος Σέλ και εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε και αγαπητά μέλη της Επιτροπής για την πρόσκλησή σας. Ε, είναι αδύνατον βέβαια να απαντήσει κανείς ε, σε τόσο ενδιαφέροντα αλλά και διαφορετικά θέματα. Πάντως αυτό είναι επί το διακύβευμα, δηλαδή δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει ας πούμε μια τέτοια συζήτηση στη Ρωσία. Τέρμα και τελεία. Αδύνατον. Δεν λέω με αυτό, δεν θέλω να ισχυριστώ ότι στη Ρωσία δεν υπάρχουν από, από άνθρωποι που έχουν διαφορετική άποψη. Υπάρχουν, αλλά η δυνατότητά τους να την εκφράσουν είτε ε, μέσα σε ένα κοινοβούλιο, είτε σε ΜΚΟ ή μέσα από ε, τηλεοπτικές πλατφόρμες ή την τηλεόραση υπάρχει μία μόνο ε, ένα κανάλι εθνικής εμβέλειας που αυτό όμως ε, ε, μπορεί κανείς ε, να το παρακολουθήσει μόνο μέσα από το διαδίκτυο. Η Ρωσία βεβαίως έχει ξεπεράσει τη Γερμανία όσον αφορά την ευρυζωνικότητα. Πραγματικά η Ρωσία έχει γίνει υπερδύναμη στην ευρυζωνικότητα και αυτό είναι επικίνδυνο για την κοινωνία και για τον έξω κόσμο. Το δεύτερο λοιπόν που θέλω να επισημάνω είναι ότι αυτά όλα είναι μέρος του προβλήματος. Δηλαδή μην κάνετε λάθος. Ε, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι δεν είναι ότι κατά κάποιον τρόπο εξεντανικεύουμε ό,τι συμβαίνει στις κοινωνίες μας. Όχι, δεν το κάνουμε αυτό και εμείς ε, είμαστε αυτοί που είμαστε. Ε, το ΝΑΤΟ έχει και αυτό τις ε, δυσκολίες του. Παρόλα αυτά, για να προχωρήσει κανείς ένα βήμα πιο πέρα και να προσπαθήσει να προσφέρει κάποια ποιότητα, θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Αν ας πούμε το νομικό σύστημα της Ρωσίας άξιζε τον κόπο έστω το όνομά του, τότε γιατί η πλειοψηφία των Ρώσων επιχειρηματιών ούτε καν ασχολούνται με το να καταφύγουν στη δικαιοσύνη στη Ρωσία. Γιατί πάνε στο Ρότερνταμ και σε άλλα μέρη. Με άλλα λόγια, το όλο θέμα δεν είναι ότι έχει να κάνει με ένα είδος DNA, πέσε το πως θέλετε, της ρωσικής κοινωνίας. Όχι κάθε άλλο είναι ότι η κοινωνία βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση και σας είπα προηγουμένως η κοινωνία είναι το πρώτο θύμα της προπαγάνδας. Το θέμα είναι το εξής, εφόσον τα γνωρίζουμε όλα αυτά, όλα αυτά έχουν και επιχειρησιακές προεκτάσεις. Είναι σαν να ε, βάζει κανείς μπροστά μας ένα καθρέφτη και οι απαντήσεις που θα δώσουμε θα πούν πολλά και για μας τους ίδιους. Με άλλα λόγια, εναπόκειται σε εμά το πώ θα απαντήσουμε. Ε, σε ορισμένα πράγματα μπορούμε να επιλέξουμε να μην απαντήσουμε γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Αλλά στη τελική ανάλυση, και εδώ μιλάω εξ ονόματος του ΝΑΤΟ, σε τελική ανάλυση δεν μπορούμε να ξεχνάμε την ε, αδυσόπιτη, μόνιμη, ε, κατάσταση, προπαγάνδα, χωρίς σεβασμό έναντι άλλων ε, κρατών, έναντι άλλων απόψεων. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι ότι μπορούμε όλα αυτά να τα γνώμε, γιατί έχουν συνέπειες, πρέπει να αντιδράσουμε σε όλα αυτά και πάλι σας επαναλαμβάνω, δεν θα αντιδράσουμε με τη δική μας την ε, προπαγάνδα, ε, δεν θα καταπιέσουμε την ε, πλειοψηφία των απόψεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και τέλος, ο ψυχρός πόλεμος. Αυτός δεν είναι όρος που χρησιμοποιούμε εμείς. Εμείς θέλουμε το διάλογο στη Ρωσία. Και έχουμε διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Έχουμε συναντήσεις ε, όπου επιθυμούμε να γίνονται πιο πολλά. Το πρόβλημα είναι ότι από την άλλη πλευρά ε, χρησιμοποιείται όρος ψυχρός πόλεμος. Πρόσφατα τον χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός Μεντέντιεφ. Δεν τον χρησιμοποίησαμε εμείς και αυτό παρακαλώ να το έχετε κατά νου. Ακόμα και αν θέλετε να επικρίνετε τις προσπάθειές μας, βεβαίως και είστε ε, ευπρόσδεκτοι στο να το κάνετε, αλλά σας λέω ορισμένα πράγματα μην τα βάζετε στο ίδιο καζάνι. Γιατί υπάρχουν πολλοί στη Ρωσία που δεν είναι ευχαριστημένοι με την κατάσταση και για αυτούς θα είναι κακό. Θα πιστέψουν ότι κάτι πάει καλά και με τις δικές μας αξίες. Γιατί σε τελική ανάλυση η αλήθεια είναι μόνο μία και τουλάχιστον κανονικά δύο και δύο κάνει τέσσερα. Η κυρία Μακόνεν. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις. Σε τρεις πτυχές θα εστιάσω. Καταρχήν ότι η ρωσική προπαγάνδα ισχύει και για την Ανατολική Ευρώπη και για την υπόλοιπη Ευρώπη και τη ΣΥΠΑ και όλο τον κόσμο. Δηλαδή δεν θα πρέπει να το περιορίσουμε μόνο στις όμορες με τη Ρωσία χώρες. Έχουμε την περίπτωση του Σιλοβιάνσκ και την ε, άλλη τη γερμανική περίπτωση που ε, αφορούν τη μία άκρη της Ευρώπης η μία και την άλλη άλλη. Υπάρχει και το Russia Today. Αν καταλαβαίνει κάποιος αγγλικά, ε, γερμανικά, ρωσικά, αραβικά και μια ακόμη γλώσσα μπορεί να διαβάσει. Μάλλον να ακούσει αυτό το κανάλι παντού και έτσι να ενημερωθεί εντός αγωγικών όπου και αν είναι. Το άλλο είναι τι μπορούμε να κάνουμε και αν πρέπει κάτι να κάνουμε. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω δύο πράγματα. Πρώτον, η δυνατότητα αντίδρασής μας είναι περιορισμένη. Δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό που κάνει η Ρωσία, όπως είπε και ο συνάδελφος, ούτε και θέλουμε να το κάνουμε, γιατί έχουμε τις αξίες μας και τις αρχές μας, ε, ε, τις οποίες θέλουμε να διατηρήσουμε. Μας είναι προσφυλής η ελευθερία μετακίνησης, η ελευθερία λόγου, τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε κατ' εμέ θα ήταν να εξηγήσουμε, να εκπαιδεύσουμε, να πούμε ποιες είναι οι αξίες μας ε, στον κόσμο για να μην μπερδεύονται και να ξεχωρίζουν πότε πρόκειται για προπαγάνδα και πότε για ελευθερία λόγου. Και επίσης πρέπει να χρησιμοποιούμε στοιχεία, πραγματικά περιστατικά και όχι αυτά που δεν υπάρχουν. Και αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας και το λέω με τη θετική έννοια γιατί υπό το πρίσμα και των συζητήσεων που γίνονται για τους ε, πρόσφυγες στην Ουκρανία στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι αρχίζουν να διερωτώνται. Πρόκειται για ελευθερία διακίνησης. Μήπως θα έπρεπε την ελευθερία κάπως να την περιορίσουμε. Αλλά αυτή είναι μια από τις αξίες μας και μια από τις ελευθερίες μας και δείχνει πολύ απλά ότι πρέπει να εξηγήσουμε και να υπενθυμίσουμε στους συμπολίτε μας. Ποιες είναι αυτές οι θετικές πτυχές των τεσσάρων ελευθεριών για τις οποίες αγωνιστήκαμε. Η άλλη πτυχή αφορά ε, την εκπαίδευση πάντα, αλλά την εκπαίδευση των συμπολιτών μας στο να μπορούν να κατανοήσουν και να μην χάνονται μέσα σε αυτή την τεράστια σφαίρα πληροφόρησης ψηφιακής εποχής. Ίσως ήδη από τα παιδιά στο σχολείο πρέπει να ξεκινήσουμε. Πού πρέπει να ψάχνουν ε, πληροφορίες, πώς να τις αναλύουν, πώς να αναζητούν ε, τα πραγματικά γεγονότα, πώς να ρωτάνε ερωτήσεις. Και αυτό αφορά και τους δημοσιογράφους Είπατε ότι κάποιες φορές, ναι, αναπαράγονται τα ε, γεγονότα. Το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε στον τύπο των χωρών μας και εμείς. Άρα θα πρέπει ίσως και αυτό να μας απασχολήσει, να δούμε πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε στις νέες αυτές συνθήκες, στη νέα εποχή των πληροφοριών, την νέα ψηφιακή εποχή που ζούμε όπου οι πληροφορίες έρχονται με τεράστια ταχύτητα και οι δημοσιογράφοι θέλουν να βγάλουν ε, πάρα πολύ γρήγορα το ρεπορτάζ και τους ενδιαφέρει μόνο να φύγει γρήγορα το ρεπορτάζ. Υπάρχει αυτή, αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ ε, των δημοσιογράφων. Δεν αρκεί όμως η ταχύτητα, πρέπει να διατηρήσουν οι δημοσιογράφοι τον επαγγελματισμό τους και οι πληροφορίες ε, έχουν αξία. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τα τρία μέλη του πάνελ για την εξαιρετική τους δουλειά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου που έλαβαν το λόγο σε αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση. Θα σας παρακαλέσω ωστόσο να παραμείνετε γιατί ακολουθεί αμέσως το επόμενο και μάλιστα δύο είναι τα επόμενα σημεία πολύ σημαντικά. Η πρώτη ε, έκθεση είναι μια έκθεση δύο πρωτοβουλίας αλλά επιτρέψατε μου πρώτα να χαιρετήσω τους προσκεκλημένους μας.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 really big and so. Okay, so let me know if we can assist. Ladies and gentlemen, please. Καθίστε παρακαλώ κυρίες και κύριοι. Το επόμενο σημείο της διάταξης είναι η πρώτη εξέταση του σχεδίου έκθεσης για τις διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα. Συγητής είναι ο κύριος Μπόκταν Σντρογεύσκη, Απολωνός από το ΕΛΚ. Η γνωμοδότηση της ΙΤΡΕ θα συνταχθεί από τον κύριο Μαρινέσκου. Και οι δύο συγητές είναι παρόντες, τους καλωσορίζω. Νομίζω είναι εδώ και περισσότεροι σκιώδη. Έχουν αποφασιστεί μάλλον ποιοι θα είναι. Προθεσμή των τροπολογιών 23 Φεβρουαρίου, ώρα 12 το μεσημέρι, όπω και στι προηγούμενε εκθέσει. που συζητήθηκαν χθε. Να μην καθυστερούμε άλλο όμω να δώσω το λόγο αυτή αμέσω στον εισηγητή κύριο Σντρογεύσκη. Pani Przewodnicząca, zacznę od podziękowań dla, dla Pani Przewodniczącej za wprowadzenie. Καταρχάς ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε γιατί έχετε εδώ και καιρό προωθήσει αυτό το θέμα. Είναι η πρώτη φορά που τα δορυφορικά συστήματα αντιμετωπίζονται με τόσο ενδιαφέρον στην Επιτροπή ΣΕΝΤΕ. Δεν θα σας αναγνώσω το σύνολο της έκθεσης. Να σας πω απλά ότι οι διαστημικές τεχνολογίες, οι δορυφορικές τεχνολογίες και οι εξελίξεις σε αυτούς τους τομείς αποτελούν προϋπόθεση για την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την τεχνολογική πλευρά αλλά και από την πλευρά της άμυνας και της ασφάλειας. Σε μια εποχή όπου αναπτύσσονται οι διαστημικές τεχνολογίες νομίζω ότι και εμείς ε, μπορούμε να ε, δώσουμε τη δέουσα προσοχή για να βελτιώσουμε τις οικονομίες, μας, ε, τις οικονομίες των χωρών μας. Έχουμε το Κοπέρνικους και το Γκαλιλαίο, τα δύο αυτά συστήματα που όμως διαφέρουν πολύ μεταξύ τους και σε ό,τι αφορά την ύψος της των δορυφόρων και σε ό,τι αφορά τον κύκλο ζωής των δορυφόρων και σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα και τα επίπεδα ε, πρόοδου, δηλαδή το πόσο προηγμένα συστήματα χρησιμοποιούν, τον καλό GPS, είναι μια εναλλακτική προς το αμερικανικό GPS σύστημα. Το καλλιλέο όμως θα δημιουργηθεί κατά τρόπο έτσι, ώστε να είναι πιο ακριβή τα δεδομένα και με μικρότερα ποσοστά σφάλματος. Το Κοπέρνικους, πολύ γρήγορα τώρα, είναι ένα σύστημα παρακολούθησης ε, γεωδεσικών πληροφοριών ε, θα μπορεί να ανταποκρίνεται ίσως και σε κλιματικές αλλαγές, παρακολουθεί τις αλλαγές του κλίματος. Ποιο είναι τώρα το βασικό καθήκον, αν θέλετε, αυτών των δορυφορικών συστημάτων, να βοηθούν τις υπηρεσίες των, των κυβερνήσεων κρατικές υπηρεσίες, μεταφορές συγκοινωνίες, πρόβλεψη πρόγνωση καιρού, καταπολέμηση τρομοκρατίας, ενεργειακή ασφάλεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν όμως και για ακαδημαϊκούς σκοπούς, ανθρωπιστική βοήθεια και ανταπόκριση σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Τι απαιτήσει προβλέπονται για αυτά τα project. Πρώτα απ' όλα, οικονομικές εγγύησεις, μεγαλύτερη προβολή, PR, πιο ενοποιημένη, πιο ενιαία γραμμή ε, στην Ένωση επίσης σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Τώρα, έρχομαι στην έκθεσή μου. Θα είδατε αναμφίβολα ότι έχω κάποιες λέξεις κλειδιά, γεωργία, κλίμα, ενέργεια, τρομοκρατία, εξωτερικά σύνορα, κρίση και άλλους σχετικούς όρους, όρους πολύ σημαντικούς και πρόκειται άλλωστε για αλληλεξαρτώμενα μεταξύ τους θέματα. Συζητούμε πολύ πρόσφατα το σχέδιο Juncker στο Κοινοβούλιο. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας όμως ότι το σχέδιο Juncker πρόκειται, αφορά επενδύσεις που θέλουν να αυξήσουν την οικονομική και χρηματοπιστωτική μόχλευση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το 2014 80 δισεκατομμύρια ευρώ σιωρευτικά απανήθηκαν σε όλο τον κόσμο για την τορυφορική τεχνολογία. 80 δισεκατομμύρια. Και τα κέρδη ήταν 151 δισεκατομμύρια. Άρα ακόμη και αν δεν έχουμε μόχλευση, έχουμε τετραπλάσια επιστροφή της επένδυσης. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επένδυση και θέλω να τονίσω για μια ακόμη φορά το πόσο μεγάλη σημασία έχει η ανάπτυξη των δορυφορικών τεχνολογιών. Σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα για διαστημικές εφαρμογές, εφαρμογές σχετικές με το Κοπένικος και το Γκαλιλαίο, για την ασφάλεια. Εδώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη δορυφορικές επικοινωνίες, ηλεκτρονικές πληροφορίες, ανταλλαγή πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που διακρίνει τις ευρωπαϊκές τεχνολογίες από τις ρωσικές, αμερικανικές, κινέζικες κτλ. είναι ότι είναι το μόνο μη στρατιωτικό σύστημα, το μόνο σύστημα που δεν το έχουν φτιάξει στρατιωτικοί για στρατιωτικούς σκοπούς κατά κύριο λόγο. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι το δορυφορικό σύστημα των ΗΠΑ είναι αποκλειστικό στρατιωτικό. Ούτε σημαίνει ότι μόνο όσες δυνάμεις έχουν την ε, δέουσα κρατική στήριξη ε, θα μπορούν να συμμετέχουν. ιδιωτικές εταιρείε συμμετέχουν και αυτές στις δορυφορικές τεχνολογίες για να προωθήσουν τα εταιρικά εμπορικά του συμφέροντα. Το ίδιο ισχύει και για την Ευρώπη. Έχουμε νεοειδριόμενες εταιρείε το 2014 το 25% των νεοειδριόμενων ήταν ε, ιδιωτικές για τον τομέα αυτό. την έκθεση μου αναφέρω και κάποιες συστάσεις αλλά και κάποιες απλές ιδέες για το μέλλον. Στις συστάσεις αυτές γίνεται λόγος για την ανάγκη καλύτερης χρήσης των διαθέσιμων πόρων και μέσων. Μιλάμε για 11 δισεκατομμύρια, δεν και λίγα. Θα πρότεινα λοιπόν αυτά τα χρήματα να τα χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε το δίκτυο ασφαλείας στην ε, Ευρώπη. Πρόκειται, επαναλαμβάνω, για μη στρατιωτικό σύστημα δορυφορικό που θα μπορούσε όμως να αξιοποιηθεί και για την υποστήριξη του αμυντικού μας συστήματος. Δημιουργήθηκε ως εναλλακτικό ε, σύστημα απέναντι σε άλλα συστήματα, να μας βοηθήσει να μειώσουμε την εξάρτησή μας από άλλα συστήματα. Παραδείγματος χάρη το GPS, τον είπα, και να μας καταστήσει πιο αυτόνομους. Δεν θέλω όμως να ε, περιστούμε στις λεπτομέρειες τώρα. Ε, εσείς μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση, να δείτε όλα τα στοιχεία. Να αναφέρω όμως ότι οι ιδιοφορικές τεχνολογίες, οι διαστημικές τεχνολογίες αποτελούν προϋπόθεση για την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Για την Επιτροπή μας όμως, και αυτό είναι σημαντικό ε, επίσης, είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα. Ευχαριστώ. Κύριος Μαρινέσκου, από πλευράς Επιτροπή Σύντρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χρειάζεται η ΚΕΠΑ την ε, δορυφορική τεχνολογία. Θέση, εντοπισμός, εικόνα, επικοινωνία και με τον Κοπέρνικο και με τον Γαλιλαίο θα πρέπει να καθαριστεί τι πρέπει να γίνει ούτως ώστε να μπορέσουν τα συστήματα να εξυπηρετούν την ε, ΚΕΠΑ. Στο γης μέλλον σε μόλις λίγους μήνες θα έχει γίνει αυτό. Και έτσι θα δημορφεί το μέλλον των συστημάτων. Τώρα όσον αφορά την επικοινωνία θα πρέπει να διαλέξουμε. Να επιλέξουμε μεταξύ εναλλακτικών. Αναβάθμιση σήμερα δυνατοτήτων η υιοθέτηση νέων συστημάτων για την Ευρώπη. Ίσως συνδυασμός αυτών των δύο εναλλακτικών. Πρέπει βέβαια και κάποια οικονομική αξιολόγηση να εξασφαλιστούν ποιοτικές υπηρεσίες και να εντοπιστεί ποιες είναι οι ανάγκες ε, και για πολιτικούς και για στρατικούς σκόπους. Ευχαριστώ κύριε Φροντζούλικα που είναι ο σκιώδης εισηγητής για τους σοσιαλδημοκράτες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι. Συμφωνώ 100% με την εισήγηση ότι δηλαδή θα πρέπει να αναβαθμίσουμε τις διαστημικές δυνατότητες για ασφαλεία και άμυνα. Αυτό σε, σε κλίμακα παγκόσμια και αυτό είναι επιθυμητό και είναι και αναγκαίο. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει τέτοιε δυνατότητες για το διάστημα. Το συντομότερο δυνατό. Είναι πάρα πολύ βασικό να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα σημερινά προβλήματα σε ασφαλεία και άμυνα. Και ε, επίσης στην εκθεσή μα θα πρέπει να αναφέρουμε όλη την ποικιλία ε, περιπτώσεων που χρειάζεται αυτό για τι απειλέ. Δηλαδή χρειάζονται οι δορυφόροι πληροφόρηση, και και θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα αν θέλουμε να μπορούμε να καλύψουμε τις μελλοντικές ανάγκες και να θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε σχέση με τους άλλους όπως την Ρωσία ή την Κίνα. Όπως ξέρετε κυρίες και κύριοι υπάρχουν κάποιες χώρες που θεωρούν ότι η κυριαρχία στο μέλλον και η επιτυχής ε, διενέργεια πολέμου εξαρτάται από αυτές τις διαστημικές δυνατότητες. Άρα θα πρέπει κανείς να έχει διαστημικά όπλα. Άρα θα πρέπει να γίνει σχετική έρευνα. Έχει γίνει επομένως μια πραγματική κούρσα, ένας αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στο διάστημα όπου η κυκλοφορία πυκνώνει και θα πρέπει να δούμε τι άλλες επιχειρησιακές δυνατότητες ε, μπορούμε να αποκτήσουμε για να έχουμε πιο ισχυρό ρόλο και άρα θα πρέπει να δούμε βέβαια το να μην έχουμε στρατιωτικοποίηση του διαστήματος. Θα πρέπει να συνεργαστούμε όσο γίνεται περισσότερο στα διεθνή φόρα και έτσι να προλάβουμε να μην ακολουθήσουν αυτή την οδό της στρατιωτικοποίησης και άλλοι στο μέλλον. Εν θα σας πω ότι συμφωνώ να έχουμε περισσότερη συνεργασία με τις ΕΠΑ όσον αφορά αυτές τις διαστημικές δυνατότητες να συνεργαστούμε και με τους Ιάπωνες αλλά και με τον ΝΑΤΟ για αυτές τις δυνατότητες και να προσπαθήσουμε να μην υπάρξει επικάλυψη των δικών μας δυνατότητων με αυτές του ΝΑΤΟ. Τελευταίο αλλά σημαντικό. Συγχαρητήρια στον ε, συγητιστή. Δεν σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα για τους ευθέρους ο κύριος Νικολάη. Κυρία. Οι διαστημικές δυνατότητες είναι το θέμα μας ε, και μπορούμε αυτές τις ε, δυνατότητες να τις ε, χρησιμοποιήσουμε και σε άλλους τομείς όπως τη διαχείριση των συνόρων, στη θαλάσσια ασφάλεια, στη γεωργία, κλιματική αλλαγή, ενεργειακή ασφάλεια, ανθρωπιστική βοήθεια και διαχείριση κρίσεων. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης, διαστημικής παρακολούθησης ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει βέβαια να προχωρήσει και σε θέματα σχετικής τεχνολογίας. Εμείς πιστεύουμε ότι ο διαστημικός τομέας θα πρέπει να είναι προτεραιότητα της ε, νέας ε, στρατηγικής και εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε υπέρ της πολιτικής, ε, μη στρατιωτικής δυνατότητας δηλαδή, αλλά και ενδεχομένω η στρατιωτική στον τομέα της ε, άμυνας και της ασφάλειας, τα κράτη-μέλη πρέπει να συμμετέχουν ε, σε διμερείς πρωτοβουλίες, να προσπαθήσουν να οργανώσουν κοινά προγράμματα και επίσης πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη, να βρούμε ε, να εμπνευστούμε από τη στρατηγική των Αμερικανών. Εξάλλου να υπάρχει και στενή συνεργασία ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να είναι προτεραιότητά μας. Αναμφίβολα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο του συστήματος Κοπέρνικος και Γαλιλαίος αυτών των συστημάτων, αλλά πιστεύουμε επίσης ότι είναι απολύτως απαραίτητο να συνεχίσουμε να στηρίζουμε διαστημικούς οργανισμούς όπως ε, τα ευρωπαϊκά συστήματα διαστημικής πλοήγησης. Οφείλουμε να γνωρίζουμε ε, και το θέμα της ιδιωτικοποίησης του διαστημικού τομέα. Αυτό πρέπει να παραμείνει. Βεβαίως χρειαζόμαστε ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα, διαστημικό πρόγραμμα για λόγους άμυνας και θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η διπλή χρήση αυτών των ε, δυνατοτήτων. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η οικονομική υποστήριξη είναι τεράστια, και η τρέχουσα οικονομική κατάσταση ε, δεν είναι βέβαια και η καλύτερη για υποστήριξη. Τέλος, θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εκδώσει μια λευκή βίβλο για την ασφάλεια και την άμυνα, διότι ως έχουν τα πράγματα, ε, ως έχουν οι εξελίξεις στην ε, αμυντική πολιτική, χρειαζόμαστε να προβάλλουμε το δικό μας το όραμα ε, στο πλαίσιο μιας λευκής βίβλου. Και θα υπάρξουν τροπολογίες, αλλά σε γενικές γραμμές στηρίζουμε το σχέδιο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Λόζινγκ είναι σκιώδη συγγήτρια. Παρακαλώ, έχετε το λόγο αυτό το σχέδιο της έκθεσης ε, για τις ε, διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την άμυνα. Ε, σε αυτήν θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλές παράγραφοι με τις οποίες δεν συμφωνούμε. Εμείς θέλουμε να υπάρχει καθαρά μη στρατιωτική χρήση του διαστήματος και των διαστημικών δυνατοτήτων. Αναφέρομαι κυρίως στις παραγράφους ε, του σχεδίου και παραθέτω η Ευρωπαϊκή Ένωση να προάγει τη συνεργασία και το συντονισμό με το ΝΑΤΟ τέλος της ε, παράθεσης. Και πέρα από αυτό υπάρχει πρόθεση τις διαστημικές δυνατότητες να τις χρησιμοποιήσουμε για τη διεξαγωγή πολέμου και παραθέτω και πάλι να φτάσουμε μέχρι τη διαχείριση κρίσεων ε, και ε, μέχρι και πραγματικές πολεμικές επιχειρήσεις. Θεωρούμε ότι σε όλα τα διαστημικά προγράμματα ευθύς εξ αρχής ε, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα προαπαιτούμενα αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 11. Επίσης, εκεί που γίνεται λόγος για ε, διαστημική τεχνολογία με διτό τομέα χρήσης για την ανάπτυξη της ε, Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Εξοπλισμών, παράγραφος 18, και εκεί είμαστε επιφυλακτικοί. Και θα ήθελα να σας επισημάνω ότι μεταξύ άλλων υπάρχει το πρόγραμμα Κοπέρνικος και Γαλιλαίος ε, τα οποία ε, χρηματοδοτούνται από μη στρατιωτικά κονδύλια. Και εάν όμως αυτά τα ε, συστήματα χρηματοδοτούνται, χρησιμοποιούνται γενικότερα. Αυτό σημαίνει ότι απορρέουν από τον κοινοτικό προπολογισμό, άρα δηλαδή παραβιάζεται το άρθρο 41.2 της συνθήκης. Και για το λόγο αυτό δεν στηρίζουμε την έκθεση, θα καταθέσουμε τροπολογίες και μπορεί να χρειαστεί να καταθέσουμε και τη δική μας έκθεση. Δεν ξέρω ε, κατά πόσον ε, ο εισηγητής θέλει να απαντήσει στα σχόλια των σκιωδών θα ήθελα να απαντήσω σε όλα αυτά που είναι πολύ σημαντικά για μένα. Και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μαρνέσκου για τη δουλειά που έκανε. Ε, οι επικοδομητικές παρατηρήσεις ενισχύουν την, έκθεση. Είναι παρατηρήσεις που μπορούν να ε, χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα. Επίσης, θα ήθελα να απαντήσω και σε αυτή την τελευταία πρόταση. Ε, πάρα πολύ προσεκτικός στην εκθεσή μου, στην ορολογία που χρησιμοποίησα. Μιλάω για δορυφόρους ε, που χρησιμοποιούν για ε, στρατιωτικούς σκοπούς. Εγώ μιλάω για την ασφάλεια πολύ γενικά. Η ασφάλεια ε, περιλαμβάνει την κλιματική αλλαγή, τις εθνικές τις θεομηνίες, αλλά περιλαμβάνει και συγκεκριμένες τεχνολογίες για να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατία χωρίς, ε, αν δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία της ασφάλειας, τα δορυφορικά συστήματα δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπίσουμε κυβερνοεπιθέσεις. Οι ε, απειλές ε, που υπάρχουν στην Ευρώπη δεν είναι μόνο τρομακρατικές αλλά και άλλες φύσεις, δεν μπορούμε να τις ε, αγνοούμε το όλο σύστημα ε, θα συνεχίσει να χρηματοδοτείται ως χρηματοδοτείται μέχρι τώρα. Εγώ δεν ζητάω να υπάρξει αλλαγή της ε, βασικής χρηματοδότησης, αλλά θα ήθελα να προσθέσω και το ότι η ανάπτυξη της διαστημικής τεχνολογίας θα κρίνει κατά πόσον η Ευρώπη και οι πολίτες είναι ασφαλείς ε, ή όχι. Κύριο Στάραν έχει ζητήσει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πάρα πολύ γρήγορα για να ρίξω κάποιες ε, πράσινες σκιές. Είμαι και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που δεν μας ικανοποιούν ε, και τα οποία ίσως τυχαίως δεν τα αναφέρετε στην εκθεσή σας. Ό,τι αφορά τα οικονομικά ε, που χρησιμοποιούνται, τους πόρους που χρησιμοποιούνται για το Γαλιλαίο, ο προϋπολογισμός έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τον αρχικό, που ήταν 5 δις και έχει φτάσει ήδη στα 13 δις. Άρα, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι δύσκολο να επιχειρηματολογήσουμε ότι κάθε ευρώ που επενδύουμε στην διαστημική τεχνολογία ε, έχει επιστροφή. Και σε ό,τι αφορά το οικονομικό κόστος, συμφωνώ και εγώ ότι υπάρχει δυνατότητα συγκέντρωση κοινή χρήση, που and share, και ελέγχου του κατά πόσο γίνεται σωστή χρήση των δημοσίων οικονομικών, αλλά υπάρχει το εξή δίλημα. Αν θέλουμε να έχουμε ωφέλη για την ΚΕΠΑ, θα έπρεπε να δούμε στο σκέλος του προπολισμού μήπως θα μπορούσαμε να διαθέσουμε κάποια από τα κονδύλια του προπολισμού προ την επίτευξη αυτών των στόχων από τα κονδύλια που έχουμε στο πλαίσιο της ε, κοινή πολιτικής ε, ασφάλειας και άμυνας. Τελευταία παρατήρηση. Σωστά αναφέρεται ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την αξιοπιστία των υφιστάμενων συστημάτων. Δεν καταλαβαίνω πολύ καλά πώς μπορούμε να πείσουμε την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου, για παράδειγμα, αυτές τις επενδύσεις να τις δει ως μεγαλύτερη προτεραιότητα σε σχέση με αυτά που συζητούμε. Παραδείγματος χάρη, τα απαραίτητα χρήματα πρέπει να δοθούν για τη διαχείριση της μεταναστευτικής και της προσφυγικής κρίσης. Ξέρουμε ότι γίνεται μια σχετική συζήτηση παράλληλα σε μια άλλη αίθουσα. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες. Θα να δούμε πώς θα επεξεργαστούμε αυτά τα θέματα και υπάρχει και κάτι ακόμη. Ο, μια ιδεαλιστική και αισιόδοξη άποψη είναι όλα αυτά τα απόβλητα τα διαστημικά που υπάρχουν και κινούνται γύρω-γύρω από τον πλανήτη μας, πώς θα μπορούσαμε να τα ξεφορτωθούμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ενημερώθηκα ότι υπάρχει και ένα ακόμη μέλος από την Επιτροπή Ήτρε που θα ήθελε το λόγο. Η κυρία Βάνιου Χόιζερ, κάπως έτσι, θέλετε το λόγο. Oh. No. Okay. Όχι. Czy pan poseł Zdrojewski chciałby odnieść się do tej ostatniej uwagi? Mi postele te και sikita, na να te katy akomi. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε το σημείο αυτό. Να σας πω τώρα την προθεσμία για τις τροπολογίες που έκτηκε την 23η Φεβρουαρίου. This day. το μεσημέρι. Next point of our agenda. Τώρα το επόμενο σημείο σημείο στις τάξεις. Εδώ έχουμε την τιμή να παρίσταται ο Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, ο κύριος Γιώχαν Ντίτριχ ε, Βέρνερ. Καλώς ορίσατε, λέει η πρόεδρος. Α, και κάτι άλλο ενημερωτικό. Η αντιπροσωπεία μας θα κάνει μια αποστολή στο Νόρδεικ τον ε, Μάρτιο. Και πρόκειται να έχουμε μια μακρά προπαρασκευή για ε, να ολοκληρώσουμε τη σημαντική έκθεση για τις διαστημικές δυνατότητες. Και τώρα χωρίς άλλη χρονοτριβή, καλώς όρισε ο κύριος ε, Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαστήματος, ο κύριος Βέρνερ. Το θέμα μας είναι να ανταλλάξουμε απόψεις με τον κύριο Γενικό σε σχέση με την δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής διαστημικών δυνατήτων για ασφάλεια και άμυνα. Σύμφωνα και με όσα ακούσαμε από την ε, εισήγηση του κ. Στριεύσκη. Είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε επομένω τι ε, εξελίξει στον τομέα αυτό. Και τώρα έχει κοιτάξει τον κύριο Βένερ για να μα ε, παρουσιάσει την εισήγησή του. Έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ, σα ευχαριστώ που μου δώσατε για την ευκαιρία να σα μιλήσω για το διάστημα σε σχέση με άμυνα και ασφάλεια. επίση είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεσή σα Μπράβο στους ε, εισηγητές Ντρογεύσκη και Μαρινέσκου. Ξέρετε, Βεβαίω ε, γινόμαστε μάρτυρες ε, μεγάλων αλλαγών. Μιλήσατε για την επικοινωνία, μιλήσατε για τις άλλες προλήψεις και είναι σαφές ότι όλα αυτά αποτερούν κάποιες προκλήσεις που πάνε πολύ περιπέρα από ασφάλεια και άμυνα. Όμως θα πρέπει να λάβουμε τα πάντα υπόψη. Επομένως πρόκειται τώρα για μια παρουσίαση ευρύτατη ε, που ξεκινά όμως με τα θέματα της ασφάλειας. Και μιλώντας για ασφάλεια έχουμε κάποια βασικά θέματα όπως ε, την ελευθερία, την άμυνα, την ασφάλεια κλπ. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά έχουν ένα κοινό στοιχείο. Ποιο είναι αυτό ότι όλα αυτά γίνονται σεβαστά και αναγνωρίζονται και επισημένονται μόνο όταν υπάρχει έλλειμμα, όταν μας λείπουν, όταν δεν τα έχουμε. Οπότε κανείς δεν δίνει δεκάρα για όλα αυτά όταν αυτά είναι εξασφαλισμένα. Και γι' αυτό είναι σημαντικό, ιδίως σε πολιτικό επίπεδο, να ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι πτυχές, ακόμα και όταν δεν μας λείπουν. Πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και ταυτόχρονα θα πρέπει κανείς να δει τι γίνεται στην κοινωνία, τι γίνεται στη βιομηχανία και στην πολιτική για τις παγκόσμιες προκλήσεις, αλλά και για τις προκλήσεις της ασφαλείας. Οπότε εμείς θεωρούμε ότι στο διάστημα πρέπει να βρούμε ένα εργαλείο, ένα εργαλείο για να καλύψει όλες αυτές τις πτυχές που είπαμε. Γεωργία, θαλάσσια πολιτική, μεταφορά, ενέργεια, ε, βιομηχανία, αλλά βέβαια και για εξωτερική πολιτική, για ασφάλεια και άμυνα. Επομένως, το διάστημα τώρα δεν είναι μόνο ζήτημα κύρου, Είναι εργαλείο άσκηση πολιτικής. Επομένως, υπάρχει πάρα πολύ στενή σχέση μεταξύ όλων αυτών των επιμέρους πτυχών του θέματος. Να δούμε τι έχει αλλάξει, τι χρειάζεται να γίνει. Ε, έχουμε τις, τους περιφερειακούς πολέμους, έχουμε την ε, πειρατεία, έχουμε τις ασύμετρες αναμετρήσεις, έχουμε ε, τις μεγάλες καταστροφές, Έχουμε το θέμα της διατροφικής ασφάλειας, τη μετανάστευση, οπότε και η ασφάλεια είναι κάτι ευρύτατο. Βεβαίως και ξεκινά με το θέμα παρατήρησης και επικοινωνίας. Η πλοήγηση ήδη αναφέρθηκε, είπαμε για τον Γαλιλαίο, για τις κρατικά λεγόμενες δημοκρατίες, για τις υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά επίσης ξαναγυρίζω είναι και το θέμα της ρύθμισης της κυκλοφορία στο διάστημα. Στο μέλλον θα είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό, αλλά βέβαια και η κυκλοφορία, παρακολούθηση και επίση η ασφάλεια αυτή τώρα αφορά ε, διαφορετικές και διαφορετικά ζητήματα. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα ε, πώς θα να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, γιατί έχουμε το Horizon 2020 που αφορά και την έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για την ε, έρευνα στον τομέα της ε, άμυνας. Βλέπετε εδώ έναν ολόκληρο κατάλογο από ζητήματα, ακόμα δηλαδή και το ζήτημα του χάρτη της μετανάστευσης που καταρτίζεται. Οπότε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος ήδη διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην δημιουργία ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής δυνατοτήτων που αφορά βέβαια και ασφάλεια και άμυνα να δούμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων στο διάστημα ή από το διάστημα. Ήδη αναφέρθηκε τι γίνεται στο διάστημα. Είπαμε ότι έχουμε σωρό φόρους, οπότε θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδου τροχέα του διαστήματος, ούτως ώστε να ρυθμιστεί το ζήτημα των δορυφόρων. Και από το διάστημα μπορεί κανείς να παρατηρεί την γη. Αυτό αφορά την ασφάλεια κατά θάλασσα, έλεγχο συνόρων, γεωργία, ε, θεομηνίες και μετανάστευση. Ο Κοπέρνικος επίσης αναφέρθηκε το σχετικό πρόγραμμα της Ένωσης. Συμβάλαμε και εμείς σε αυτό τα διάφορα domains για τις εφαρμογές. Είπαμε ότι θα ισχύσει και κατά θάλασσα. Και με τον Κοπέρνικο γνώση έχουμε ένα εργαλείο το οποίο δεν αφορά μόνο κάποιους δορυφόρους αλλά χρησιμοποιεί δεδομένα επιτόπου χρησιμοποιείται και από αέρος. Και έτσι έχουμε όλο αυτό το αμάλγαμα δεδομένων, ούτως ώστε τελικά να μπορεί κανείς να έχει τα δεδομένα που χρειάζονται για να λάβει αποφάσεις. Τώρα από πλευρά τη ασφάλεια στη θάλασσα. Σημαντικό. Έχουμε πρώτα πρώτο θέμα της ε, πειρατείας, έχουμε τους λιμένες, την ε, πλοήγηση μεγαλών πλοίων. Χρειάζονται πάρα πολύ τα συστήματα πλοήγηση επομένω, γιατί ακόμα και το καλύτερο σήμα του Γαλιλαίου δεν αρκεί. Χρειάζεται ένα αναβαθμισμένο σύστημα που να είναι προσαρμοσμένο στις τοπικές ανάγκες, γιατί θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια και ακρίβεια κάτω από 10 εκατοστά. Επομένω χρειάζεται και η σχετική επιμελητία, προστασία για την θαλάσσια ασφάλεια. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται με τις δραστηριότητε των πειρατών. Είμαι σίγουρο ότι θα γνωρίζετε τι γίνεται με το σύστημα αυτόματου εντοπισμού. Μπορούμε από το διάστημα να εντοπίσουμε πλοία. Να το συγκρίνουμε με το σήμα της ISAT με οπτικούς αισθητήρε. Και αν υπάρχει κάποια απόκληση, τότε πάει κάτι στραβά με το πλοίο και θα ξαναεξετάσουμε τα πράγματα. Αν δείτε λίγο αυτή την εικόνα, θα διαπιστώσετε ότι στην Βαλτική θάλασσα, στην Βόρεια θάλασσα, τόσο κοντά δηλαδή σε εμά, δεν εμφαίνονται πλοία. Αυτό δεν ισχύει. Υπάρχουν τόσα πολλά που δεν μπορεί ο εντοπισμός να τα βρει και να δώσει πληροφορίες. Όμως να βλέπουμε ότι οι δορυφόροι έχουν κάποιο είδους τηλεσκόπιο, τηλεσκόπιο κυμάτων, ούτω ώστε να μπορούν να ελέγξουν τέτοιου είδους ε, περιοχές όπως η Βαλτική ή η Βόρεια Θάλασσα. Πριν από κάποια χρόνια συγκροτήθηκε ο χάρτης του διαστήματο για να καλύψουν τι θεομηνίες όπως ας πούμε ε, σεισμούς, ε, δασοπυρκαγιές και όλοι όσοι προσυπέγραψαν ε, συμμετέχουν πλήρως. Να βλέπετε τώρα το τσουνάμι της Ιαπωνίας. Έχει ενεργοποιηθεί από τους προσφογράψαντες το σύστημα, υπάρχουν οι πληροφορίες και συλλέγονται επομένω όλα τα δεδομένα ούτω ώστε να μπορεί κανείς να βοηθήσει όπου χρειάζεται και να δει τι χρειάζεται να γίνει αναφέραμε την μετανάστευση. Αλλά και εδώ το διάστημα βοηθάμε κάποιες εφαρμογές. Βλέπουμε τις ροές των μεταναστών, τα στρατόπεδα, τα σύνορα. Αν δείτε όμως αυτή την ε, λίστα δραστηριοτήτων θα δείτε και άλλα. Θα δείτε τι μπορεί να υποστηριχθεί από το διάστημα. Και έτσι είναι εφικτό κάποιος να μην μετακινηθεί παρά τις οικονομικές δυνατότητες. Πώς μπορεί να αναπτύξει κανείς την πατρίδα του αντί να μεταναστεύσει. Βλέπουμε επομένως τι γίνεται με την ξηρασία, βοηθάμε στην ε, ίδρευση, την παιδεία, ε, την έμπνευση τελικά γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι θα πρέπει ο κόσμος να είναι εμπνευσμένο και στις χώρες εκείνες όπου τώρα η κατάσταση είναι τραγική. Να τους έρθει η έμπνευση να μείνουν και βλέπουμε ότι βοηθά το διάστημα. Εξού και αυτός ο χάρτης διαστήματος και μεταναστευσής. Τώρα, θέματα ασφάλειας. Είναι η χρήση της διαστημικής τεχνολογίας και του τέφλων το οποίο φυσικά δεν είναι διαστημικό υλικό, αλλά έχει σχέση. Βλέπετε λοιπόν εδώ αριστερά αυτό που τώρα έχει γίνει φαινόμενο συχνό στην Ευρώπη, αυτές τις μεγάλες ουρές κόσμο που περιμένει μία ουρά για να ελεγχθεί, να μπορεί να πάει κάποιο όπερα από ουρά για να μπω στο κοινοβούλιο. Είχαμε όμως την ε, τεχνολογία να μπορούμε να κάνουμε έλεγχο άμεσα χωρίς ε, άλλου είδους ιδιαίτερες συσκευές. Οπότε ελέγχουμε τον κόσμο καθώς περπατάμε σε ένα ε, κτίριο. Αυτό χωρίς ακτινοβολία. Ελέγχουμε την ακτινοβολία που έχει το σώμα γιατί όλοι έχουμε κάποια ακτινοβολία και είναι αρκετά ισχυρή, ούτω ώστε να μπορούμε να δούμε τι γίνεται. Όλα αυτά αφορούν την, ε, ε, την τεχνολογία και την διαστημική. Ε, Επίση, μπορούμε να δούμε τις κινήσεις του πλήθους ε, σε κάποιες εκδηλώσεις βλέπουμε όταν υπάρχει ε, μετακίνηση, κάποιοι τρέχουν και έτσι δίνουμε πληροφορίες στην αστυνομία και σε άλλες αρχές για να υπάρξει ασφάλεια επίσης. Εδώ έχουμε κάποιο άλλου είδους ε, παρακολούθηση των στρατοπέδων εκπαίδευση των τρομοκρατών, τόσο να μπορούμε να κάνουμε κάτι πριν επιτεθούν. Κάτι άλλο που αφορά την αεροπορία είναι το MH370. Κρίμα είναι όταν δεν μπορεί κανείς να εντοπίσει πού ακριβώς βρίσκεται ένα αεροπλάνο. Γιατί υπάρχει τεχνολογία, αλλά δεν υπάρχουν δορυφόροι που το κάνουν. Και βλέπετε ότι δεν είναι ε, σαφές πάντα που έχει γίνει ε, η πτώση ενός αεροπλάνο, άρα μπορούμε με κάποιες αισθητήρε να βρούμε που βρίσκεται. Εκτός από τους άλλους αισθητήρε έχουμε και τον ε, δέκτη ADSB, γιατί υπάρχουν κάτι τέτοια σήματα που εκπέμπονται και έτσι μπορούμε να εντοπίσουμε το πού βρίσκεται ένα αεροπλάνο ένα πάσα στιγμή. Όμως, ακόμα δεν υπάρχουν αρκετοί δορυφόροι ή αρκετοί δέκτες σε τροχιά, οπότε ε, μπορούμε μέσα σε ένα λεπτό ή άντε σε μια ώρα να ξέρουμε τι απέγινε αεροπλάνο και πού βρίσκεται. Αν δεν έχουμε αρκετά κοντά ένα δορυφόρο. Όμω ε, υπάρχει κάπου στόλο, μπορεί αυτό να γίνει. Τώρα επειδή όσον αφορά την διαχείριση τη κυκλοφορία στο διάστημα, βλέπω εδώ πέρα έχουμε 6.000 ε, μόρια, σωματίδια τέλο πάντων, σε ένα ε, κυβικό εκατοστό στο διάστημα. Αυτό είναι κίνδυνο για του δορυφόρου. Ε, υπάρχουν και δορυφόροι που είναι εκτός ελέγχου, αλλά ξέρετε ότι πολλές φορές είναι τέτοια κατάσταση που έχουμε κάποια ε, κοσμικά σώματα που μας πλησιάζουν να εδώ βέβαια στο Τσελιαμπίνσκ ε, τι έγινε και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αποφύγουμε παρομοίες καταστροφές. Τώρα υπάρχει επίσης η έννοια της προστασίας των κρισίμων των σημαντικών υποδομών έχουμε τις ε, συνήθεις ε, λύσεις αλλά θα πρέπει κανείς να μπορεί να προλάβει το κακό και να μπορέσει μετά να διαχειριστεί την κρίση. Εδώ βλέπετε σε αυτόν τον κύκλο το τι πρέπει να ληφθεί υπόψη ούτως ώστε να έχουμε κάποιο είδου αηφόρο, βιώσιμη δραστηριότητα για ασφάλεια και άμυνα. Οπότε βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, η ΙΖΑ, ε, αναπτύσσεται τέτοιου είδους έννοιες έχει τέτοιε ιδέε που ε, καταρτίζουμε συμφωνίε με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε ένα παγκόσμιο δίκτυο όπως ε, ε, αναφέρθηκε. Έχουν πλησιάσει τους Άπωνε στενέ σχέσεις και με τους Αμερικανού με την NASA. Επίσης, έχουν αναπτύξει σχέσεις και δίκτυο με όλους όσους ασχολούνται με το διάστημα. Έχουμε εκπαιδευμένο προσωπικό που μπορούν να κάνουν ότι απαιτείται. Έχουμε και εμείς εσωτερικό σύστημα ασφάλειας, πολύ σημαντικό όταν μιλά κανείς για ασφάλεια και άμυνα. <clears throat> Έχουμε επομένω τις απαραίτητες τεχνολογίες και, και στο Νόρδεκ υπάρχουν εγκαταστάσεις που ασχολούνται με αυτό. Επίσης έχουμε και κάποιους αρχεία για τα δεδομένα που είναι γι' αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί θα πρέπει να έχουμε αρχεία που πάνε στο παρελθόν για να ξέρουμε τι υπήρχε πριν και τι έχουμε τώρα. Και τέλος, ε, γιατί άλλο το πήγαμε και είναι οι αποστολέ. Οπότε η υπηρεσία διαστήματο μπορεί να γίνει ένας ε, αρχιτέκτονας και ένα εμπειρογνώμων για την αμήνα στην Ευρώπη. Οπότε το πολιτικό μήνυμα είναι ότι είμαι 60 έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάντοτε ονειρευόμαστε τι Ηνωμένε Πολιτείε τη Ευρώπη. Ξέρω ότι αυτός ο στόχο τώρα έχει κάπω απομακρυνθεί, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι το να έχουμε ένα Ηνωμένο διάστημα για την Ευρώπη. Γιατί όλοι οι παίκτε, η Υπηρεσία Άμυνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι άλλοι εμπλεκόμενοι, όλα τα δεσμικά όργανα τώρα συνεργάζονται και οπότε μπορούμε να συνεργαστούμε προς χάρη ε, των ε, φορολογουμένων αλλά και για να πετύχουμε ασφάλεια στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Γενική. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφό μας ε, αν έχει να κάνει κάποια σχόλια. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. όλα αυτά που αναφέρθηκαν ε, τα αξιολογούμε στην έκθεση. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε εκείνους ε, που θεωρούν ότι η επέκταση είναι το κλειδί στην επιτυχία της ε, Ευρώπης. Εγώ στηρίζω τις δραστηριότητες του οργανισμού, αλλά έχω μία ερώτηση για μία παρεξήγηση που υπάρχει. Έχω λάβει την πληροφορία ότι το κόστος του προγράμματος Γαλιλαίος αυξάνεται. Βεβαίως ε, ε, αυτό μπορεί να συνέβη, αλλά υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο υλικό κόστος αφενός και στις ε, πληροφορίες που μας δίδονται. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για πάνω από 11 δις ευρώ, αλλά άκουσα πληροφορίες ότι Μέχρι τώρα το κόστος είναι 13 δις. Ε, κύριε Χόιζεν από την Ήτρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Μπέρνερ που ήρθατε σήμερα εδώ και ευχαριστούμε που μας παρουσιάσατε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν και που έχει να προσφέρει και το διάστημα. Πράγματι έχετε δίκιο με όλα τα στοιχεία που ε, μπορείτε να αποκτήσετε από το διάστημα γιατί πολλοί σκεφτούν το διάστημα είναι ένα νέο χρυσοροχείο εγώ θέλω να σας κάνω μία ερώτηση σχετικά με τη διτή χρήση διότι σε ορισμένες χώρες, ε, παραδείγματος χάρη στην Κίνα ή στις Ηνωμένε Πολιτείε, δεν υπάρχει ουσιαστικό διαχωρισμός. Βρίσκονται όλα στα ίδια χέρια και εδώ στο πρόγραμμα Κοπέρνικος έχουμε την δυνατότητα ε, να γίνεται πλήρης ε, χρήση βάση ε, όλων των δεδομένων, αλλά αυτό πάλι παρεμβαίνει ε, με το θέμα της ασφάλειας. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ, κατά τη γνώμη σας, η Ευρώπη πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το διαχωρισμό ανάμεσα στην άμυνα και την ασφάλεια φενός και αφετέρου ε, στο ότι θέλουμε να κάνουμε όσο δυνατόν πιο εμπορική χρήση των δεδομένων. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει κάποια, κάποιο ξύμορο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εχθές ε, μπορέσαμε ε, να φιλοξενήσουμε τον πρέσβη της Ιαπωνίας και τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Ιαπωνικών Ιαπωνικών Υποθέσεων που μας παρουσίασαν ε, την ε, νομοθεσία, την Ιαπωνέζικη νομοθεσία για την ασφάλεια και την ε, ειρήνη. Αναφέρθηκε η συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ιαπωνία, κυρίως στο διάστημα. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες ε, εκτόξευσης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω ότι είναι μια ερώτηση παγίδα, αλλά επειδή έχουν προκύψει πολλές περιπτώσεις ε, όπου η εκτόξευση ε, δορυφόρων δεν ήταν αυτονόητη, θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν κάποια σχέδια να συνεργαστείτε με τους Ιάπωνες ομολόγους. Μήπως Μπορείτε να μας απαντήσετε από αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Καταρχήν, όσον αφορά το κόστος του προγράμματος Γαλιλαίος, θέλω να σας πω ότι δυστυχώς ε, τα στοιχεία που αναφέρατε δεν είναι τα τελικά. Γιατί, αν το δείτε λίγα εξωστά, ε, το πρόγραμμα Γαλιλαίος είναι μόνιμη δραστηριότητα. Το GPS ξεκίνησε την δεκαετία του 60 και οι Αμερικανοί εξακολουθούν να επενδύουν στο πρόγραμμα. Δεν μπορεί δηλαδή να πει κανείς ότι εγκαθιστά ένα πρόγραμμα και μετά τελείωσε. Ε, για το πρόγραμμα Γαλιλαίος χρειάζεται κανείς ε, δορυφόρο. Ε, οι δορυφόροι έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής στο διάστημα. Όλοι λοιπόν ήδη έχουμε αρχίσει να σκεφτόμαστε για την επόμενη και τη μεθεπόμενη γενιά δορυφόρων. Ε, γιατί η επόμενη θα είναι περίπου ίδια, αλλά όσον αφορά τη μεθεπόμενη, ε, νομίζω θα θέλουμε να έχουμε ακόμα πιο εξελιγμένους δορυφόρους. Τα στοιχεία λοιπόν που αναφέρετε πρέπει να τα προσδιορίσουμε και χρονικά. Και μετά, αν θέλετε, μπορώ και εγώ να σας αναφέρω ορισμένα στοιχεία. Μετά, ε, κατηδίαν, αν θέλετε, ε, μπορώ να σας ε, πω περισσότερα στοιχεία για το θέμα το χρόνου, του χρόνου. Όσον αφορά τη διτή χρήση, ευχαριστώ πολύ και για αυτή την ερώτηση. Κοιτάξτε, για μένα προσωπικά η ασφάλεια και η άμυνα είναι μη στρατιωτικές δραστηριότητε. Είναι για να ε, προσφέρουμε ασφάλεια στην κοινωνία μας. Δεν είναι για να διεξάγουμε πόλεμο. Κατόπιν τούτου, βεβαίως οτιδήποτε αναπτύσσει κανείς, δηλαδή η τεχνολογία, ε, μπορεί να το ε, χρησιμοποιήσει και αρνητικά και θετικά. Εμείς από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος είμαστε πάντα πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε τα προϊόντα μας να χρησιμοποιούνται για ειρηνικούς σκοπούς. Αλλά και να το πω κιόλας, η ειρήνη για μένα είναι ειρηνικός σκοπός, άρα δηλαδή στη σύμβασή μας αναφέρεται ο ελληνικό σκοπό αλλά και η αποφάση του Συμβουλίου ε, σχετικά με την ειρήνη. Τώρα, όσον αφορά την ερώτησή σας για το ξύμορο σχετικά με την ανοιχτή πρόσβαση, θέλω να σας πω ότι η ανοιχτή πρόσβαση είναι περιορισμένη. Άρα δηλαδή δεν είναι ότι όλα τα δεδομένα που έχουμε τα δίνουμε ε, δωρεάν σε όλους, αλλά τα δεδομένα που έχουμε από το πρόγραμμα Κοπέρνικος και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ε, θεμητός ανταγωνισμός ε, και σε επίπεδο βιομηχανίας. Άρα δηλαδή εγώ είμαι υπέρ της ανοιχτής ε, πρόσβασης, αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτά δεν αντιφάσκουν με την ειρηνική χρήση. Όπως αφορά και στο θέμα του Γαλλαίου έχουμε ε, τα ανοιχτά και τα κλειστά, τις ανοιχτά, ανοιχτές και κλειστές υπηρεσίες. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι η χρήση για μη ειρηνικούς σκοπούς ε, αυτή θα πρέπει να είναι περιορισμένη. Η τρίτη ερώτηση αφορά στην αυτόνομη πρόσβαση στο διάστημα. Εγώ ως μηχανικός ε, θέλω να σας πω ότι το να μπορεί κανείς να κάνει κάτι αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Το να μπορεί να έχει δύο δυνατότητες αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Εμείς έχουμε κάνει μετρήσεις ε, ασφάλειας. Βεβαίως και μπορούμε να συνεργαστούμε με τους Ιάπωνες για την εκτόξευση δορυφόρων και με Αμερικανούς και αυτή τη στιγμή, μάλιστα μόλις πριν από δύο μέρες, ε, εκτοξεύουμε και ρώσικους πυράβλους. Μπορεί κανείς να το κάνει αυτό. Αλλά το να υπάρχει ευρωπαϊκή αυτονομία, αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία, γιατί σε περίοδους κρίσης ε, θα πρέπει κανείς να μπορεί να το κάνει αυτό και όταν άλλες ε, χώρες προσπαθούν να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα και εσύ δεν είσαι εκτός παιχνιδιού. Έχουμε τώρα μια νέα οικογένεια ε, που εκτοξεύουν πυράβλους είναι 62-64 ε, είναι πολύ πιο σε αυτές πλέον οι δυνατότητες ε, Θέλουμε να υπάρξει περιορισμός του κόστους περίπου το 50% για τη νέα γενιά δορυφάρων. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην αγορά και να διασφαλίσουμε την αυτόνομη πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διάστημα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ακόμα και κατά διάρκεια κρίσεων. Ευχαριστώ κυρία Γιάλα Σέντερ για το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Μας έδωσε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Έχω ένα ερώτημα. Στην έκθεση του κυρίου Σντρογεύσκη, όπως είναι φυσικό, υπάρχει και μία παράγραφος για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Θα ήθελα να μου πείτε αυτή η σχέση πώς λειτουργεί και να μου πείτε την άποψή σας και για την συνεργασία. Γιατί φαντάζομαι υπάρχουν κάποια ισχυρά ε, σήμερα και κάποιοι κίνδυνοι, θα ήθελα να μου πείτε περισσότερα. Επιστρέψαμε μόλις από την ε, UNAV4MED, που είναι το στρατηγείο της στη Ρώμη. Θα ήθελα να μου πείτε και για το ε, δορυφορικό σύστημα αν υπάρχει ένα ειδικό τμήμα για την ε, παροχή δορυφορικής υποστήριξης ε, σε καινοτόμες ε, επιχειρήσεις σαν αυτή την UNAV4. Και τέλος, είπατε ότι είναι η δορυφόροι. Πάντοτε συζητάμε και με τον Καλλιλά, αλλά δυστυχώς και με όλα τα άλλα τα ευρωπαϊκά project συζητάμε τον προϋπολογισμό και δεν συμφωνούμε. Δυστυχώς. Θα πρέπει όμως να είμαστε πιο φιλόδοξοι, αλλά τέλος πάντων, ερώτηση. Με αυτή τη νέα γενιά εκτοξευτήρων, τι θεωρείτε ότι είναι το βέλτιστο δυνατό για να αντιμετωπίσουμε τις φιλοδοξίες μιας νέας στρατηγικής κοινής στρατηγικής ευρωπαϊκής άμυνας. Thank you, madam. Ευχαριστώ. Και Γενική Διευθυντά, να έχετε την καλοσύνη να απαντήσετε παρακαλώ. Μάλιστα, πρώτα απ' όλα, Ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ. Ε, για να είμαι πολιτικά ορθός, δεν επί στη δική μου αρμοδιότητα. Είμαι επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, ενός διακυβερνητικού οργανισμού που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βέβαια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έχουμε συμφωνίες και, με, και για την χώρα και άλλες. Για το Κοπέρνικο, στον Καλιλαίο. Οπότε αυτό τον καιρό γενικώ ναι. προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να περάσουμε σε μια νέα, σε μια ευρωπαϊκή πολιτική και στρατηγική για το διάστημα. Αν έχουμε από διαφορετικά όργανα διαφορετικές στρατηγικές ε, θα έχουμε πρόβλημα. Καλό είναι να έχουμε μια νέα στρατηγική και πολιτική γιατί αλλιώς ε, τα προβλήματα που θα προκύψουν θα είναι αρκετά σημαντικά. Εμείς έχουμε καλή σχέση με την Κομισιόν, κυρίως με την Κομισιόν και ελπίζω, γιατί αυτή είναι, αυτή είναι το θεσμικό με το οποίο έχουμε κυρίως σχέση. Για τον ΝΑΤΟ δεν θα αναφερθώ και τη σχέση μας. Τώρα αναφερθήκατε στο τι μπορούμε να παράσχουμε να προσφέρουμε φυσικά την εμπειρία μας στον τομέα της πλοήγησης, επιτήρησης αεροπορικής, αλλά και στον τομέα των επικοινωνιών. Υπάρχει συζήτηση, για παράδειγμα, για ένα δορυφορικό πρόγραμμα για ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, GovSapcom λέγεται αυτό το πρόγραμμα και βέβαια είμαστε έτοιμοι να σας προσφέρουμε την τεχνογνωσία μας για την ανάπτυξη του προγράμματο αυτού σε συνεργασία πάντα με την Κομισιόν. Αυτή είναι καλή ιδέα. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά ζητήματα, τον προπολογισμό, είναι διαφορετικέ οι πηγέ. Πρώτον, κράτη-μέλη. Για κάποια συγκεκριμένη περίοδο έχουμε χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη που συνδέεται συνήθως άμεσα με συγκεκριμένα project. Και τώρα έχουμε μια επιπλέον συνεισφορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά πρέπει να έχετε υπόψη σας πώς λειτουργούν όλα αυτά. Αν τα κράτη-μέλη του ΕΖΑ έχουμε 22 στην την Ελβετία στην τη Σουηδία, στην την Ορβηγία, συγγνώμη, αυτά τα κράτη μας δίνουν χρήματα και θέτουν κάποιες υψηλές απαιτήσεις, ε, high level requirements τις λέμε εμείς. πρέπει να εφαρμόσουμε, να εκτελέσουμε ε, αυτές τις τάσεις. Το ίδιο ισχύει με την Κομισιόν. Η Κομισιόν είναι αυτή που ορίζει αυτές τις high level requirements και εμείς είμαστε αρχιτέκτονες ε, που θα πρέπει να χαράξουμε ε, το πρόγραμμα, τις τεχνολογίες του πτυχές σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση που με ρωτήσατε, εν μέρη προέρχεται από την ε, Ένωση και την Κομισιόν και εν μέρη από τα κράτη-μέλη. Πάντοτε προσπαθούμε να υποβάλουμε προτάσεις για προγράμματα που θα μπορούσαν να υποστηριχθούν άμεσα από τα κράτη-μέλη. Δεν μπορώ να ζητώ χρήματα και να κάνω μετά ό,τι μου αρέσει εμένα. Αυτοί είναι οι κανόνες που έχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Πάντοτε λοιπόν οι αποφάσεις λαμβάνονται σε σχέση στενή με τα προγράμματα και τα project. Ευχαριστώ. Ο, η Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γενική Διευθυντά για τις πληρέστατες πληροφορίες που μας δώσατε και για τις απαντήσεις σας και τις παρατηρήσεις σας. Να προσθέσω κάτι ακόμη, έτσι, για να καταλάβετε κάπως το κλίμα. Στην Ευρώπη τα χρήματα για το διάστημα ε, αντιστοιχούν σε 10 λίτρα βενζίνης για κάθε Ευρωπαίο πολίτη αναχρόνο. Άρα κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα πλήρωνε 10 ε, λίτρα βενζίνης ε, το χρόνο, θα δίνει ένα ποσό. Αυτό το ποσό αντιστοιχεί ε, σε εμά. δεν είναι και τόσα πολλά. Μάλιστα, καλό μάρκετινγκ κάνατε, καλό μάρκετινγκ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ και βασιζόμαστε και στην περαιτέρω συνεργασία, περαιτέρω επαφές θα γίνει θα στείλουμε και αντιπροσωπεία ε, της ε, υποεπιτροπής μας. Στο Nordic, την έδρα σας. Σας ευχαριστούμε και τώρα πάμε στα διάφορα. Αν δεν υπάρχουν διάφορα, σας ενημερώνω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας είναι στις 3 Μαρτίου λύεται η συνεδρία. Σας ευχαριστώ.